Madame la Présidente Linda, mes chers collègues. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, προτείνω να επανέλθουμε στις εργασίες της Επιτροπής ΤΑΞ 2 και να κηρύξουμε την άναξη αυτή της κοινή συνάντηση της Επιτροπής Ανάπτυξης. Γι' αυτό και χαιρετίζω εδώ την παρουσία της Πρόεδρου της ε, Λίδα Μακάβεν και των μελών της και της Επιτροπής ΤΑΞ 2. Η συνεδρίαση αυτή είναι αφιερωμένη στις συνέπειες του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Με τη Λίδα Ματκάβεν λοιπόν θελήσαμε να έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις, να έχουμε αυτή την ακρόαση, γι' αυτό και ευχαριστώ όλες τις προσωπικότητες που δέχτηκαν έρθουν και να προσφέρουν τις μαρτυρίες του Θελήσαμε λοιπόν να έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων σε μια στιγμή όπου διάφορες εργασίες, διάφορες αποκαλύψεις, δημοσιογραφικές, άλλες ακροάσεις που έχουν γίνει εδώ υπό την πρωτοβουλία της ΤΑΞ 2 και όχι, στα Εθνικά Κοινοβούλια, στον Νοσά και αλλού. Όλα αυτά λοιπόν έδειξαν αφενός μεν το μέγεθος της φοροαποφυγής, από την οποία εποφελούνται διάφορες μεγάλες πολυεθνικές και από την άλλη μεριά τις συνέπειες, τις οικονομικές και πολιτικές συνέπειες αυτού του φαινομένου της φοροαποφυγής σε πολλές χώρες. Αδικίες σε όλες τις χώρες μέλη, αλλά οι συνέπειες είναι ακόμα πιο μεγάλες παγκοσμίως. Γι' αυτό λοιπόν και σκεφτήκαμε ότι είναι σημαντικό πριν να ολοκληρωθούν οι εργασίες της Επιτροπής Τάξη και δεδομένων των προτεραιοτήτων της ε, Επιτροπής Ανάπτυξης να μπορέσουμε να συναντηθούμε για δύο ώρες εδώ στις Βρυξέλλες. Δεν ε, θα πω περισσότερα. Θα δώσω το λόγο ευθύ αμέσω στην Λίντα Μακκάβεν με την οποία από κοινού θα προεδρεύσουμε σήμερα. Λίντα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαμασούρ. Είναι πολύ σημαντικό πράγματι να συνεργαστούν οι επιτροπές μας πάνω σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα της φορολογίας. Για αυτούς που δεν εργάζονται με την ανάπτυξη, ίσως να γνωρίζουν ότι το Σεπτέμβριο που μας πέρασε η διεθνή κοινότητα πέρασε στο επόμενο στάδιο της ε, αναπτυξιακής συνεργασίας για να επιτευθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι του 2030. Ε, Συγχρόνω στην Αντή Αβέμπα, τον Ιούλιο που μα πέρασε, υπήρξε μια άλλη διάσκεψη στην οποία η διεθνή κοινότητα είπε θέλουμε ανάπτυξη για τα επόμενα 15 χρόνια και θέλουμε να την πετύχουμε. Ναι, σίγουρα η αναπτυξιακή βοήθεια είναι σημαντική, ο ιδιωτικό τομέας είναι σημαντικός, αλλά ο, η μεγαλύτερη πηγή πρέπει να είναι η κινητοποίηση των ενδογενών πόρων. Αυτή είναι η στόχη λοιπόν για τα επόμενα 15 χρόνια. Όταν όμως ακούμε ότι πολλές αναπτυσσόμενες χώρες δυσκολεύονται να εισπράξουν φόρους επειδή είτε πιέζονται από τις πολυεθνικές προκειμένου αυτές να συνεργαστούν, ζητούν ε, χαμηλούς ε, φόρους, τους υπόσχονται δηλαδή ότι θα πληρώσουν χαμηλούς φόρους ή επειδή υπάρχουν ε, παράνομες ροές χρημάτων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη που φεύγουν από τη χώρα και καταλήγουν σε λογαριασμούς, σε φορολογικούς παραδείσους, όχι μόνο στον Παναμά, αλλά και στο Λονδίνο και αλλού. Τότε λοιπόν λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε μεταξύ μας για να μην συμβαίνει αυτό. Γιατί δεν μπορείς να φτιάξεις μια αξιοπρεπή κοινωνία, δεν μπορείς να έχεις αξιοπρεπείς υπηρεσίες αν δεν καταπολεμήσεις την φοροποφυγή. Πρέπει να είναι κανείς σίγουρος ότι τα χρήματα αυτά από τους φόρους εισπράττονται αφενός και αφετέρου χρηματοδοτούν υπηρεσίες ποιότητας. Έτσι λοιπόν σήμερα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε πριν από τη διάσκεψη της Αντίς Αμπέμπα τι γίνεται με την φοροποφυγή στις αναπτυσσόμενες χώρες. Όμως δεν χρειαζόμαστε πια λόγια, χρειαζόμαστε δράση κύριε Λαμασούρ και ξέρω ότι εσείς είστε αποφασισμένος η χώρα σας να αλλα... η χώρα σας, συγγνώμη, η επιτροπή σας να αλλάξει την ε, κατάσταση. Και όσα κάνει καλή δουλειά, αλλά τώρα χρειάζεται μια νέα όθηση. Ο κόσμος αυτό περιμένει, έχει βαρεθεί να ακούει για αυτά τα προβλήματα και να μην βλέπει λύσει. Γιατί όλοι λένε ναι, πρέπει να κάνουμε κάτι, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Χρόνο το χρόνο δεν βλέπουμε αποτελέσματα. Λίγοι τελικά ξέρουμε ότι υποφελούνται πολύ, αλλά και πολλοί πληρώνουν για αυτούς οι οποίοι υποφελούνται. Θα έχουμε δύο πάνελ ειδικών. Θέλουμε να ξέρουμε τι γίνεται τώρα και τι θα κάνουμε. Χαίρομαι λοιπόν που έχουμε μαζί μας τον κύριο Στεφάνο Μανσερβίση που είναι ο νέος διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης στην ΤΕΦΚΟ ξέρω ότι υπάρχει μια μικρή μονάδα η οποία δουλεύει πάνω στα φορολογικά. Τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορείτε να φροντίσετε να έχετε τη συνεργασία που χρειάζεται για να φέρετε αποτελέσματα όσον αφορά τα φορολογικά αυτά ζητήματα και την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Ναι, Ευχαριστούμε για την πρόσκλησή σας. Έχουμε βρεθεί και σε άλλες στιγμές της ε, επαγγελματικής μας ζωής. Πρέπει να ξέρετε ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα πώς οι γενικές διευθύνσεις συνεργάζονται για να λύνουν τέτοια προβλήματα. Εδώ μιλάμε για χρηστή διακυβέρνηση, έτσι, περί αυτού πρόκειται. Το σωστό πολιτικό μείγμα είναι αυτό το οποίο μας προσφέρει προσανατολισμούς. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά και για τη σημερινή συζήτηση και για το μελλοντικό μας έργο. Γνωρίζετε, το είπατε εξάλλου, ήταν και στην καρδιά της Αντίς Αμπέμπα για τους στόχους του 2030 και το μήνυμα κλειδί που βγήκε γι' αυτό και είναι πρόκληση για μας για το μέλλον, είναι η κατάργηση της στόχιας, η εφόρος ανάπτυξη, πράγματα τα οποία δεν μπορούν να επιτεθούν παρά μόνο αν έχουν χρήματα οι χώρες και αντιμετωπίσουν δηλαδή τα οικονομικά τους και δημοσιονομικά τους ζητήματα. Είναι μια μεγάλη ευθύνη Το μέγεθος των προβλημάτων είναι τεράστιο. Οι εκτιμήσεις λένε ότι πάνω από ένα 3 δολάρια χάνεται κάθε χρόνο μέσα από παράνομα οικονομικά κανάλια. Μια Ήπειρος, όπως είναι η Αφρική, που όλοι μιλάμε για επενδύσεις, χρηστή διακυβέρνηση κτλ. 6% είναι οι απώλειες του ΑΕΠ ετησίως στην Αφρική. Γι' αυτό μιλάμε και δεν είναι λίγο. Αυτό λοιπόν πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το πάνελ υπό τον Μπέκη στην διάσκεψη αυτή πρότεινε ακριβώς συνεργασία. Κατά τη γνώμη μου, η συνεργασία είναι κάτι πολύ θετικό. Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί το ζήτημα είναι να αργαστούμε συντονισμένα. Να μην λέμε εγώ, εσύ, δεν είναι δυνατόν ο ένας να δίνει μαθήματα ηθικής στον άλλον. Όχι, πρέπει να βρούμε το σωστό μείγμα, το σωστό τρόπο. Η Επιτροπή έχει εκπονήσει ένα έγγραφο το οποίο καλύπτει αυτές τις πτυχές. Πώς θα συλλέξουμε περισσότερα χρήματα περισσότερους φόρους, πώς δηλαδή θα έχουμε μια πιο αποτελεσματική φορολογική πολιτική και ε, καλύτερες δαπάνες, που σημαίνει πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα χρήματα αυτά υπέρ της ανάπτυξης. Αυτό το Collect to More, Spend Better, αυτός είναι ο τίτλος της ε, ανακοίνωσής μας του 2010 όσον αφορά τη φορολογία και την ανάπτυξη. Και αυτό ακριβώ ήταν και η βάση Τη καλή συνεργασία που είχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Κοινοβούλιο. Δεν αρχίζουμε λοιπόν από το μηδέν. Είναι περιορισμένη η εμπειρία μας. Αλλά υπάρχει και δείχνει το μέγεθος της δέσμευσή μας υπέρ ακόμα καλύτερη συνεργασία στο μέλλον. Η συλλογή ε, περισσότερων φόρων σημαίνει αντιμετώπιση της ε, φοροαποφυγής και των παράνομων φορολογικών πρακτικών. Και στη συνέχεια το spend better, το να δαπανάμε καλύτερα, σημαίνει ότι τα χρήματα αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται για στόχους, ευγενείς στόχους, κοινοφελείς. Τώρα, θέλουμε ένα καλό παράδειγμα. Ο καθένας θα πρέπει να είναι πολύ ταπεινός. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα παράδειγμα που είναι εξαιρετικό, αλλά η προσπάθειά μας είναι να ρυθμίσουμε περισσότερο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τελευταίο πακέτο για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής έχει και μία εξωτερική πτυχή. Ακριβώς προκειμένου η ευρωπαϊκή φορολογική πολιτική να ευθυγραμμίζεται με τις αναπτυξιακές μας πολιτικές. Πολιτική συνοχή, έτσι, και ενεργός μάλιστα. Δεν ελέγχουμε μόνο απλώς, συνδυάζουμε αυτά που κάνουμε για μας με αυτά που κάνουμε για τους εταίρους μας. Πολύ σύντομα θα αρχίσουμε συζήτηση με τις χώρες μέλη και όλους τους εταίρους προκειμένου μαζί να αξιολογήσουμε την φορολογική πολιτική των χωρών μελών στα πλαίσια της αναπτυξιακής πολιτικής. Τώρα για την παγκόσμια εταιρική σχέση. Collect More, Spend Better έχει εντοπίσει 10 τομεί για την ε, βελτίωση και για την ανάπτυξη διεθνών ε, προδιαγραφών με τη συμμετοχή όλων. Γιατί εννοείται ότι όλοι πρέπει να συμμετέχουν, όλοι πρέπει να ε, θεωρούν δικό τους θέμα την υπόθεση αυτή. Με τους εταίρους λοιπόν έχουμε καταλήξει σε πρωτοβουλία για την κινητοποίηση πόρων στο εσωτερικό των χωρών και αποφυγή των φορολογικών παραδείσων για να διαχειριστεί κανείς το δημόσιο χρήμα και εκείνο τον φορολογούμενο στις αναπτυσσόμενες χώρες, αυτό είναι μια τεράστια πρόκληση, γιατί σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει χρηστή διακυβέρνηση και αυτό δεν είναι μόνο ε, θέμα ποσοτικό, έχει να κάνει και με τη λογοδοσία των αρχών απέναντι στους φορολογούμενους. Έχουν περιμένει πάρα πολλοί φορολογούμενοι σε αναπτυσσόμενες χώρες γι' αυτά. Μερικές φορές ε, τα χρήματα δίνονται μέσω αναπτυξιακής βοήθειας, ενώ εδώ θέλουμε τους πολίτες των χωρών αυτών να τους βάλουμε στο κέντρο της πολιτικής μας. Δουλεύουμε λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση. Συνεργασία, πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης 20, συνεργαζόμαστε με τον ΟΙΕ προκειμένου να ενημερώσουμε τις προσπαθειές μας με τον ΟΣΑ για να ενισχυθεί το πλαίσιό μας για συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επίσης για να υπάρχει στέρεα εταιρική σχέση για μεταφορές πόρων και όσον αφορά την διαχείριση των πόρων. Υπενθυμίζω εδώ ότι πριν από δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε μια πρωτοβουλία αντίστοιχη. Σήμερα σκεφτόμαστε και άλλους τομείς που συνδέονται ακριβώς με την προσέγγιση μας αυτή που είναι η προστιθέμενη αξία, ότι η χρηστή διακυβέρνηση είναι η προστιθέμενη αξία. Είναι και αυτό κομμάτι του παζλ πάνω στο οποίο δουλεύουμε. Και ολοκληρώνω με μεταξύ, όπως είπα και στην αρχή, εδώ δεν πρόκειται μόνο για ένα νέο τομέα που μπορούμε να αναπτύξουμε περισσότερο, αλλά είναι και ένας τρόπος για να βελτιώσουμε την παγκόσμια διακυβέρνηση. Σε συνεργασία με διάφορες γενικές διευθύνσεις θα ακολουθήσουμε την αρχή που λέει δεν θα φροντίζουμε μόνο για τους άλλους, θα φροντίζουμε για το τι κάνουμε και εμείς και τα δύο. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να χτίσουμε πάνω στα θεμέλια που έχουμε ήδη βάλει, να ενισχύσουμε την εταιρική μας σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου μαζί να βρούμε έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτό το όχι απλώς φαινόμενο, είναι κάτι πιο πολύ από φαινόμενο, το οποίο διαρθρωτικά μόνο μπορεί να αντιμετωπιστεί. Μπορείτε να βασιστείτε σε εμά λοιπόν, που και εμείς ευχαρίστως να βάλουμε τη γνώση μας, την εμπειρία μας υπέρ του κοινού μας έργου που είναι η ανάπτυξη και υπέρ μιας ε, διακυβέρνησης καλύτερης και με περισσότερη διαφάνεια. Ευχαριστώ. Merci Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γενική Διευθυντά, ο Πρόεδρος, για την εισήγησή σας, η οποία ήταν ε, αρτιότατη, πληρέστατη και ε, καλό κουράγιο βέβαια για τα καινούργια σας καθήκοντα. Τώρα, ας αρχίσει η συζήτηση. Πρώτο πάνελ. Ακριβώ όπως είπε η κυρία Μακάβα, θα έχουμε δύο πάνελ. Οπότε και εγώ θα διευθύνω την συζήτηση για το πρώτο πάνελ. Θα προεδρεύσετε στο δεύτερο πάνελ η Λίντα. Για το πρώτο πάνελ, Δυστυχώ, ο κύριος ε, Ολομό, που είναι χρηματοοικονομικός επίτροπο Αφρικανικής Ένωση δεν μπόρεσε να προσέλθει και ζητήσει γνώμη διότι ασθενεί. Αλλά έχουμε τρεις προσωπικότητε. τρεις ε, ικανοτάτους οι οποίοι ήρθαν και τους ευχαριστούμε. Πρώτη η κυρία Ατίγια Βόρες, η οποία ε, διδάσκει στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου του Ναϊρόμπι και φαίνεται από το βιογραφικό της ότι επίσης έχει περάσει από άλλα πανεπιστήμια Ρουάντα, Νοτιοαφρικανική Ένωση, Βιέννη από το Lancaster University της Αγγλίας ε, από την ορδηγία κλπ. Ο κύριος Μανουέλ Μόντες, ο οποίος είναι ε, σύμβουλος ε, στο Κέντρο Οικονομικής Ανάπτυξης της Γενέβης, ο οποίος επίσης έχει διδάξει και έχει ερευνήσει σε μία σειρά χωρών. Έχει περάσει από τη Σρι Λάνκα, Φιλιππίνες, Χονολουλού, Σιγκαπούρη. Qui, après Επίσης, Στάνφορντ της Καλιφόρνια και κάτω με κύριο Ρόσφαλντο, που ήδη έχει έλθει να μας μιλήσει στην ε, Επιτροπή μας που ασχολείται ε, με την διαμόρφωση της πολιτικής ως σύμβουλος για τα θέματα τα φορολογικά και ισότητας. Εκπροσωπεί την Oxfam και έχει ασχοληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορες χώρες με αυτό το θέμα. Έχει πάει και στην Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα. Ο επίση ε, έχει διδάξει αλλά και έχει εργαστεί για τα θέματα ισότητα γυναικών ε, στο Αρμόδιο Υπουργείο της Γαλλίας. Ο κάθε ένας από τους καλεσμένους μας παρακαλούμε να μιλήσει πέντε λεπτά ούτως ώστε να εισηγηθεί το θέμα του. Και στη συνέχεια πρέπει να δώσουμε τον λόγο στους συναδέλφους με το σύστημα Eye. Κυρία Βόρης, έχετε το λόγο. Σα ε, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Είναι τιμή μου που είμαι εδώ πέρα. Θα αναφερθώ λίγο στην εξωτερική σας στρατηγική και στον αντίκτυπο που ίσως έχει ή δεν έχει στις αντσόμενες χώρες και θα αναφερθώ στην έρευνα που έχουν κάνει για την Κένια και εξετάζει το πώς επηρεάζει η φορολογική νομοθεσία πριν ξεκινήσει όλη αυτή η μεταρρυθμιστική διαδικασία και μετά. Και ένα πράγμα το οποίο παρατήρησα στην εξωτερική σας στρατηγική που αναγγείλατε τον Ιανουάριο φέτος. Μιλάτε για δίκαιο και αποτελεσματικό φόρο στις επιχειρήσεις και βεβαίω κάποια μέτρα για να αποφευχθεί η κατάχρηση. Και βεβαίως το θέμα της διαφάνειας. Οπότε το ζήτημα είναι πόσο ευρεία είναι αυτή η συζήτηση περί διακυβέρνησης και βεβαίω το ζήτημα το φορολογικό είναι πολύ ευρύτερο. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ να προσθέσω κάποια θέματα στην όλη συζήτηση. αποτελεσματικότητα είναι κάτι το οποίο ήδη αναφέρθηκε. Επίσης η δικαιοσύνη, κάτι το οποίο προκύπτει. Άκουσα ήδη την λογοδοσία από τον νέο γραμματέα και βεβαίως το θέμα της ευθύνης. Η διαφάνεια καλύπτεται και προχωρά, αλλά τα υπόλοιπα ακόμα έχουν μείνει πίσω. Οπότε, τι πρέπει να τονίσουμε. Στην προηγούμενη συζήτηση άκουσα να μιλάμε για κρατικές ενισχύσεις οι οποίες επηρεάζουν τις αναψώμενες χώρες. Χαίρομαι λοιπόν που το θίγουμε το ζήτημα και χαίρομαι που μια χώρα επίσης ε, χρηματοδοτεί με αυτή την λογική. Η λογική του να ξοδεύουμε καλύτερα και να συλλέγουμε περισσότερα, εγώ θα την έλεγα αντίστροφα. Η λογική σας μάλλον, είναι να συλλέγουμε περισσότερα και να ξοδεύουμε καλύτερα. Εγώ θα το έλεγα αντίστροφα. Γιατί πολλές αμψόμενε χώρες και στην Αφρική έχουν, έχουμε πολύ κακή πολιτική όσον αφορά τις δαπάνες. Οπότε αν μείνουμε στη συλλογή το θέμα των δαπανών ε, παραμελείται. Οπότε θα πρέπει να δούμε αυτό το ζήτημα που περιλαμβάνει και τη διαφθορά και όλα τα άλλα μη δασμολογικά εμπόδια. Και πράγματι η ατζέντα της ε, Άντις ε, Αμπεμπά τα αναφέρει αυτά. Επίσης η πλατφόρμα σας για την ορθή διακυβέρνηση είναι ενδιαφέρουσα αλλά δεν έχετε παραμέτρους. Π.χ τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μήπως υπονομεύουν την ορθή διακυβέρνηση άλλων κρατών. Και είναι κάτι το οποίο προέκυψε στην ε, συζήτηση, δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια σαφής αντίληψη των παραμέτρων αυτών και άρα ποια είναι και τα κριτήρια επιλογής και ποια κράτη στη μαύρη λίστα και ποια όχι. Επίση θα ήθελα να υπάρχει μια κατάταξη των κρατών με βάση τις ικανότητες και θα ήθελα εδώ πέρα να αναφερθώ στην Κένια. Είναι μία από τις πέντε χώρες, ε, τι οποίε θα λέγαμε χώρες μεσαίου εισοδήματο στην Αφρική, άρα είναι σε κάπω διαφορετική κατάσταση από άλλε που είναι οι ελάχιστα ανεπτυγμένε. Προσπαθούμε π.χ Προσπαθούσαμε τότε, παραδείγματο χάρη, να πάμε τη Unilever στα δικαστήρια για το transfer pricing και χάσαμε μεταξύ άλλων γιατί δεν είχαμε βάση δεδομένων, δεν είχαμε τις δυνατότητες τι εμπορικέ. Από το 2004 έχουμε πλέον τα στοιχεία της ε, εφορίας και αυτό γιατί ο ΩΣΑ εκπαίδευσε τους υπαλλήλους μας. Μετά ξεκίνησε η υπόθεση Καρουτούρη. Αυτό είναι σημαντικό γιατί δεν πρόκειτο για μια πολυεθνική του Βορρά, είναι μια πολυεθνική Ινδική, οπότε τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο περίπλοκα από ό,τι πριν. Πριν η συζήτηση αφορούσε βόρειες εταιρείε που έρχονται και κάνουν όλες αυτές τις άδικες ε, πρακτικές, αλλά τώρα υπάρχουν πολλές νότιες πολυεθνικές και από άλλες χώρες, οπότε αν δεν φτιάξουμε το σύστημα θα έχουμε όλο και περισσότερες εταιρείε που θα έρχονται και θα κάνουν αυτά τα πράγματα. Ε, από όταν λοιπόν προέκυψε η υπόθεση Καρουτούρη δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες μου από την ε, εφορία υπήρχαν και άλλες τρεις εταιρείες ε, οι οποίες όμως συμβιβάστηκαν με τις αρχές χωρίς περαιτέρω συζητήσεις. Οπότε έχουμε εδώ πέρα αντίκτυπο που περιλαμβάνει και βρετανικές εταιρείες και άλλες. Ε, δεν μπορώ να σας πω τα ονόματα όμως των υπολείπων. Επίσης ενδιαφέρον είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ε, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αλλάξει ελαφρώς ε, θέση και μας δίνει πληροφορίες, αλλά από την άλλη η Γερμανία έχει μια υπόθεση που εκκρεμεί στα δικαστήρια και μας λένε πως οι πληροφορίες τις οποίες ζητάνε οι φορολογικές αρχές είναι πέρα από την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Οπότε παρά το ότι γίνεται κάποια δουλειά στη διαφάνεια δεν αρκεί. Υπάρχουν διαφορές στο πώς οι ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν την Κένια. Οπότε, έχουμε και αφρικανικές πολυεθνικές Οπότε, ανέφερα την Ινδία, αλλά έχουμε και την Ιγυρία, την Κένια, Νότιο Αφρική και την Αίγυπτο, που έχουν πλέον πολυεθνικές εταιρείε. Οπότε μετά ο φορολογικός ανταγωνισμός παραμένει και γίνεται ακόμη πιο περίπλοκο ζήτημα. Οπότε, όταν δεν είναι σαφής η μέθοδη, ε, θα γίνουν τα πράγματα ακόμη χειρότερα. Και σε μια χώρα σαν την Κένια, το θέμα δεν είναι μόνο να λαμβάνουμε πληροφορίες, αλλά θα πρέπει και εμείς να δίνουμε. Λοιπόν, να σας πω ποια είναι τα ζητήματα τα οποία ακόμα δεν έχουν επιληθεί πέρα από αυτά που προκύπτουν από το BEPS. Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα είναι πως δεν καλύπτεται εδώ πέρα οι εξορρυκτικές βιομηχανίες και πρέπει να το πάρουμε σοβαρά. Δεύτερον, έχουμε ζητήματα ακόμα με την μεταφορά κερδών στο εξωτερικό γιατί καμιά φορά δεν ξέρουν οι φορολογικές αρχές ποια μέθοδο πρέπει να εφαρμόσουν και δεν είναι ξεκάθαρη η νόμη. Επίσης, δεν υπάρχει τίποτα στην BEPS για τις υπεργολαβίες, οπότε οι υπεργολαβίες χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο. Η Κένια είχε μια πρόσβαση στα λεγόμενα συγκρίσιμα και τώρα οι υποθέσεις που κρατούσαν 5 και 6 χρόνια επιλύονται σε 2-3 χρόνια. Βεβαίω, ακόμα είναι πολύ αυτό ο χρόνο και δεν είμαστε τόσο αποτελεσματικοί και υπάρχουν διαφορετικέ βάσει δεδομένων. Π.χ. η PWC χρησιμοποιεί μία βάση δεδομένων, οι φορολογικέ αρχέ μία άλλη και υπάρχουν διαφορέ. Έχουμε ανενεργέ εταιρείε οι οποίε αυτή τη στιγμή δεν ρυθμίζονται και υπάρχει βεβαίω και το ζήτημα των δυνατοτήτων. Πλέον δεν μιλά μόνο για τι φορολογικέ αρχέ, δεν υπάρχουν δυνατότητε στις λογιστικές εταιρείες, στη δικαιοσύνη, για τους ερευνητές φορολογικών ζητημάτων, οπότε υπάρχει γενικότερα ένα ζήτημα δυνατοτήτων και βλέπουμε να πηγαίνουμε μπρος πίσω. Αυτά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Σας ευχαριστούμε και εμείς κυρία μου. Μανουέλ Μόντες, ο δόκτωρ, έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, μεγάλη μου Καλή μου τιμή κύριε Πρόεδρε, εδώ να απευθύνομαι στην Οικονομική Επιτροπή του Κοινοβουλίου. Εργάζομαι για το South Center που ασχολείται με τις αντισώμενες χώρες, οπότε ξέρετε ότι είμαστε κάτι σαν τον ΟΣΑ, αλλά πολύ λιγότερο, είμαστε περίπου 20 έδρα η Γενέβη, γιατί ο ΟΣΑ έχει μόνο στο Παρίσι γύρω στους 2.000 υπαλλήλους αλλά ασχολούμαι με 52 χώρες ε, και όταν μπει η Νικαράγω θα είναι η 53η χώρα. Έχουν και κάτι μεγάλες χώρες όπως Κίνα, Ινδία, Βραζιλία, μικρότερες όπως το Μαλί. Αλλά ο Σάχη μόνο 34. Το πιο σημαντικό όπως θα θέλω να σας πω είναι το εξής. Από την αρχή το λέω, ότι θα να εξασφαλίσουν ότι οι αναπτυσσόμενες θα μπορούν να επιστρατεύσουν πόρους για να πετύχουν βιώσιμη ανάπτυξη και αυτό θα πρέπει να είναι προτεραιότητα για όλους. Έχουμε στο ΟΗΕ το θεματολόγιο 2030. Αυτό θα πρέπει να ισχύει για όλο τον κόσμο, θα πρέπει να την ασπαστούν όλοι παντού. Αλλά όπως είπαμε και στην αρχή, ε, ένας από τους περιορισμούς μας για να το πετύχουμε είναι το ότι αυτές οι χώρες δεν μπορούν μόνο τους να βρουν τους πόρους και αν έχουν τις επενδύσεις για υποδομές, για παιδεία, για ανάπτυξη της βιομηχανίας. Οπότε και εξαρτώνται από το εξωτερικό για τους πόρους. Μία σημαντική μελέτη έγινε στην ε, Αφρική. Το είπαμε. Για τις παράνομες ροές χρημάτων. μπορεί να τις πούμε και παράτυπες, άλλο παράτυπη, άλλο παράνομο για το λέμε έτσι, γιατί έχουμε 60% αυτών των χρηματοοικονομικών ροών που θα μπορούσαν ε, να καταλήξουν στα ταμεία των φορικών αρχών είναι νόμιμες ροές. Μιλούμε για παράνομη διακίνηση ε, προσώπων, ε, για λαθρεμπόριο, για Έχουμε όμως ε, και άλλου είδους παρατυπίες όπως παράμε τιμολογικές πολιτικές. Να όσα ε, που το έχει αναλάβει. Έχουμε ε, επίσης για τις εξαγωγές, διπλές τιμολογήσεις, ας πούμε για τον Χαλκό, γιατί ας πούμε η Ζάμπια παράγει τον χαλκό και τον εισαγεί η Ελβετία. Η Ελβετία φτιάχνει σοκολάτα αλλά δεν φτιάχνει το κακάο. Και η εισαγωγή δεν γίνεται σε νόμιμε, με νόμιμες τιμές. Και όλα αυτά ε, σύμφωνα με τον νόμο. Το θέμα είναι κάτι το οποίο είναι νόμιμο, πώ θα κηρυχθεί παράνομο με μια μεταρρύθμιση, με μια αλλαγή. Και έτσι κάποια χώρα όπω η Ζάμπια να μπορέσει να πουλήσει τον χαλκό στην παγκόσμια τιμή. Να μην το πουλάει φθηνότερα και μετά η Ελβετία να εισάγει και να βάζει ψηλότερη τιμή. Βέβαια, είναι και θέμα φορολογία στη Ζάμπια, η οποία χρειάζεται φορολογικά έξοδα. Και ο φόρος είναι ψηλότερος από ότι μια ελβετική εταιρεία που εξάγει. Άρα 60% είναι από παράτυπες ενέργειες. ότι δεν μπορεί να φορολογηθεί. Αλλά επίσης έχουμε από την Αντίσα Μπέμπα, όταν έγινε εκείνη η συνάντηση για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, το ότι υπήρξαν προτάσεις από τις ε, χώρες να αναμορφωθεί η σχετική φορολογική επιτροπή και να αναβαθμιστεί. Γιατί έχουν τρόλους αυτές τις παράνομες ροές, όλα, ε, όλα αυτά τα πρότυπα, αυτές τις ροές, τις παράνομες, παράτυπες ε, είναι αντικείμενο μόνο του ΟΣΑ, γιατί έχουμε τις 34 χώρες του ΟΣΑ, έχουμε την γραμματεία του ΟΣΑ, οπότε και θα πρέπει να ενεργεί η γραμματεία με τρόπο που να συνάδει με τις επιθυμίες αυτών των χώρων. Και μπορεί να υποβάλει ένσταση για μια ενέργεια οποιαδήποτε από τις 34 χώρες. Έχουμε επομένως τουλάχιστον 2-3 δεν τελειώνω, τελειώνω πρόεδρε. Έχουμε θέμα της ε, μετακύληση, τέλο της μετακίνησης των, των κερδών. Γιατί είναι θέμα. Το πώς θα φορολογηθεί μία πολυεθνική. Τι θα γίνει επίσης και με τον εξορρυκτικό τομέα, που σημαντικό είναι τη Ζάμπια. Άρα, αν θέλει να βοηθήσει την ε, ανάπτυξη ο ΩΣΑ θα πρέπει να επεκταθεί για το πώς οι κανόνες του ΩΣΑ θα εφαρμοστούν ευρύτερα και όχι μόνο στα πλαίσια του ΩΣΑ γιατί εκεί υπάρχει έλεγχος και υπόκειται ο ΩΣΑ στις συνστάσεις από τα μέλη του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα έχει το λόγο η κυρία Σάντονι. Ευχαριστώ πολύ θα σας ε, μιλήσω για το έργο μας σε 90 χώρες για να καταπολεμήσουμε την υποανάπτυξη. Το θέμα της φορολογίας είναι πολύ σημαντικό αν λάβει υπόψη του κανείς ακριβώς τις ανισότητες. Οι ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν μια κοινή πρόκληση. Θέλω και εγώ εδώ να προσθέσω ότι και εμείς είμαστε στην πλατφόρμα αυτή για τη φορολογία, δηλαδή να γεφυρώσουμε λίγο πολύ τις ευρωπαϊκές χώρες με τις υπονάπτυξη. Είναι πολύ χρήσιμο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συμπεριλάβει και μια εξωτερική διάσταση στο θέμα της φορολογίας. Πολύ βασικό είναι το κριτήριο της χρηστής διακυβέρνησης. Συνήθως όσοι παίρνουν πολιτικές αποφάσεις εδώ, ε, τις παίρνουν σε ένα βαθμό απόρριτου. Αυτό ισχύει για παράδειγμα, για τους φορολογικούς παρεθύσους, για τον εταιρικό φόρο. Και έτσι δεν έχουμε πάντα θεμητό ανταγωνισμό. Καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουν άλλη λύση οι χώρες μέλη, αντί να μπουν σε φορολογικούς πολέμους, καλύτερα να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν την φοροποφυγή. Γιατί αλλιώς φτάνουμε όλοι στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Και δεν το λέω εγώ αυτό, το λέει η κυρία Λαγκάρτα. Το άλλο που βλέπουμε είναι ότι κυριαρχούν τα αποτελέσματα του ΟΣΑ και των ΜΠΕΠΣ. Οι, οι αναπτυγμένες χώρες θέλουν να επιβάλλουν τα συμπεράσματα του ΟΣΑ και των ΜΠΕΠΣ στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η διαδικασία καταλόγων. Αναφερθήκαμε πριν στη μαύρη λίστα. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι τέτοιες διαδικασίες δεν είναι νέες και το βλέπετε και στην εικόνα ότι το 2000, 2001, ακόμη και το 2015 η συζήτηση γίνεται για αυτή τη μαύρη λίστα. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να εξακολουθούμε όπως παλιά δεν λέμε ότι είμαστε κατά της ιδέας ενός τέτοιου καταλόγου, μιας μαύρης λίστας, αλλά πρέπει να πρόκειται για κάτι αντικειμενικό, με διαφάνεια. Είναι χρήσιμο στην διαδικασία, αλλά τίθεται το θέμα των κριτηρίων. Ποιος μπαίνει σε αυτή τη λίστα. Πολλές αναπτυσσόμενες ε, χώρες έχουν πρακτικές για να μειώσουν την φορολογία μεγάλων επιχειρήσεων. Υπάρχουν τόσο πολλές φορολογικές πρακτικές που έχει εντοπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι χώρες, για παράδειγμα, που έχουν την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να θεωρηθούν φορολογική παράδοση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω ότι θα μπορούσε να συντονίσει τα πράγματα και αυτό θα υποστηρίξουμε στην επόμενη πλατφόρμα. Δεν πρέπει να είναι σε βάρος των αναπτυσσόμενων χωρών ένας τέτοιος κατάλογος. Να προβλέπονται κυρώσεις. Και δεν θα πρέπει μία χώρα να στοχεύουν οι ευρωπαϊκές χώρες. Εσείς θα πρέπει να μην τα βάζετε δύο φορές με τις αναπτυσσόμενες χώρες, να μην τις τιμωρείτε διπλά. Τώρα, η τωρινή διαδικασία έχει πολιτικοποιηθεί πάρα πολύ. Μια μαύρη λίστα μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο αν έχετε αντικειμενικά κριτήρια. Αν μόνο ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή, θα υποστηρίζουν τα δικά του συμφέροντα. Είναι λογικό αυτό, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και άλλη πλευρά. Ελπίζουμε λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δουλέψει ώστε να προωθήσει αντικειμενικά κριτήρια. Έπειτα πάντα θα υπάρχουν κάποιες χώρες που δεν θα θέλουν να συνεργαστούν, απρόθυμες. Μπορεί να είναι αποτελεσματική μια μαύρη λίστα μόνο αν προβλέπονται κυρώσεις. Όλες κάποιες χώρες θα θελήσουν να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους και είδαμε τι έχει γίνει με τα τελευταία σκάνδαλα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επίσης πρώτα απ' όλα να βάλει τάξη στα δικά της πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να κατηγορούνται μόνο χώρες που δεν είναι ευρωπαϊκές. Αν υπάρχει μια μαύρη λίστα, να μπει και Αμερική. Δεν το λέω εγώ αυτό. Το είπε το 2009 ο Πρωθυπουργός Γιούνκερ πολύ ενδιαφέρον να το δει κανεί. Πόσο δηλαδή πολιτικοποιημένη μπορεί να είναι μια τέτοια μαύρη λίστα. Αν θέλετε να σας δώσω το link ε, όπου αναφέρεται αυτό. Πολλά περισσότερα θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας και ιδίω να επιστήσω την προσοχή σας στο ΕΚΟΦΗΝ που θα γίνει αύριο. Αλλά καλύτερα να αφήσουμε περισσότερο χρόνο στις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ σε ευχαριστούμε πολύ σε όσους πήραν το λόγο μέχρι τώρα για τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας που ήταν πολύτιμα. Έχω να κάνω δύο σχόλια εγώ προσωπικά αυτή τη στιγμή. Πρώτα απ' όλα για το πρόβλημα της μαύρης λίστας. είναι κάτι που το συζητήσαμε και στη... πριν από λίγη ώρα. Είναι πολύ λεπτό στην πράξη αυτό το ζήτημα. Από την άλλη, είναι σαφές ότι αυτό που ονομάζουμε μη συνεργάσιμη δικαιοδοσία πρέπει να το δακτυλοδείχνουμε. Ιδιαίτερα αν πρόκειται για κάποιες μικρές ε, τροπικές ε, νήσους κτλ. Αν βέβαια είναι μια μεγάλη χώρα, είναι πιο δύσκολο. Συγχρόνως όμως, ταξιδεύοντας ανά τον κόσμο, διαπιστώνουμε ότι η έννοια του φορολογικού παραδείσου ερμηνεύεται εντελώ διαφορετικά. Στην Ουάσιγκτον η Ιρλανδία θεωρείται φορολογικός παράδεισος απλώς και μόνο εξαιτία του 12,5%. Όταν στην Αμερική είναι 35%. Θεωρείται λοιπόν υπερβολικά χαμηλό στην Ιρλανδία και γι' αυτό τη θεωρούν ε, φορολογικό παράδοσο. Ε, δεν είναι το ίδιο με τις παρθένους νήσους όμως. Κάποιοι μας είπαν ότι η εκπόνηση ενός τέτοιου καταλόγου μαύρης λίστας είναι διπλωματικός εφιάλτης. Ευχαριστώ πάντως για τις αναλύσεις σας και θα δούμε τι συμπεράσματα θα βγάλουν οι εισηγητές. Ο κύριος Κοφούρ θα μας πει τη γνώμη του. Ο κύριος Μόντες επίσης αναφέρθηκε στον ΟΣΑ. Το έργο εκεί είναι πολύ σημαντικό. Και θέλω να χαιρετήσω εδώ ακριβώ το ρόλο του ΟΣΑ, γιατί νομικά μιλώντας, όπως είπε ο κύριος Μόντες, ΟΣΑ με 34 μόνο χώρες, ο Γενικός του Γραμματέας λογοδοτεί σε αυτές τις χώρες μόνο. Και οι τοποθετήσεις του ΩΣΑ είναι τοποθετήσεις, είναι συστάσεις, έτσι, δεν είναι αποφάσεις δεσμευτικές. Ο κύριος Γκούρια λοιπόν έχει κάνει συστάσεις και γι' αυτό το θέμα της φορολόγησης των πολυεθνικών και ΩΣΑ θέλει να συμμετέχουν στο πρόγραμμα δράσης BEPS όσο γίνεται περισσότερες χώρες και χώρες δηλαδή του G20 που δεν είναι στον νόσα και αναπτυσσόμενες χώρες που δεν είναι στον νόσα. Εγώ πρότεινα στον Γενικό Γραμματέα Γκούρια να οργανώσουμε μία διακοινοβουλευτική διάσκεψη με αυτό ακριβώς το θέμα και να προσκαλέσουμε εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων όλων των χωρών που συνεισφέρουν. Είναι μια ιδέα πρόσφατη του όσα δεν υλοποιήθηκε αυτό προς το παρόν, αλλά να ξέρετε ότι είναι ένα κοινό σχέδιο που θέλουμε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όσα. Και αυτό για να διασφαλίσουμε ότι αν για ιστορικούς λόγους ο Διεθνής Οργανισμός που είναι ο καταλληλότερος, αλλά έχει μόνο 34 χώρες, δεν μπορεί μόνος του να οργανώσουμε μία μεθοδολογία που εκπρόσωποι όχι όλων των χωρών του κόσμου, αλλά εν πάση περιπτώσει των περισσότερων από όλες τις κατηγορίες και των αναπτυσσόμενων χωρών δηλαδή, να συμμετέχουν στις εργασίες. Δύο έχουν ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ δύο λεπτά ο καθένας. Ντεμάση και Άσλι Φόξ. Και μετά ο κύριο Κοφόντ θα καταλήξει σε συμπεράσματα για αυτό το πρώτο πάνελ. Φάβιο. Sorry, I'm not used uh, to be... Συγγνώμη, ε, δεν έχω συνηθίσει να μιλάω πρώτος. Οπότε με ευνηδιάσετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα αξιόλογα μας είπατε. Αυτά για τις είπα, είπε ο κύριος Γιούνκερ. Αλλά μας την μια εβδομάδα ε, ο γερουσιαστής που προεδρεύει της Αρμόδιας Επιτροπής. Ε, και τα ακούσαν φάει και, στην, ε, και, στο, και στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Δηλαδή δεν ε, συγκρατήθηκαν τα πούνε διπλωματικά. Τα είπαν στα Ράτα. Οπότε είπαμε ότι έχουμε πάρα πολλές αναπτυσσόμενες χώρες που δεν έχουν τεχνική ε, δυνατότητα για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στα προγράμματα αυτόματη ανάλυσης πληροφοριών. Εσείς τι λέτε, πόσες ε, χώρες καλύπτονται από αυτό το πρόβλημα και πόσες θεωρείτε ότι θα μπορούσε αυτό να γίνει, θα ωφελούσε να ε, κατονομάζουμε τις χώρες μία προς μία. Να δούμε ακριβώ πού υπάρχει δράση κάποιων πολυεθνικών σε αναπτυσσόμενη χώρα. Και αν υπάρξει χρόνο, θέλω να σα πω, εσεί τι μέτρα νομίζετε θα φέρουν περισσότερη διαφάνεια σε αντισώμενε χώρε. Και να κάνουμε κάτι για τα, τα χρήματα τα οποία διαφεύγουν ε, στο εξωτερικό, τι γίνεται με κάποιους ψηλά ιστάμενους που έχουν ε, τέτοια ε, δράση. Πέστε μας τι γίνεται και με το θέμα του πραγματικού δικαιούχου. ευχαριστούμε Φαμπιό Άσλη ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ να ευχαριστήσω. Ευχαριστήσω και εγώ τους ομιλητέ μα. Έχω δύο ερωτήσει για, για τον δεύτερο ομιλητή που μίλησε για το χαλκό της ε, Ζάμπιας. Και αναφέρατε πολλές φορές την διαφορά μεταξύ παρανόμων και παρατύπων, όπως είπατε, πρακτικών. Ε, με συγχωρείτε, αλλά δεν έχουν μεγάλη διαφορά, ιδιαίτερα στα αγγλικά αυτές οι λέξεις. Ε, Ειδικά οι δύο λέξεις που είπατε στα αγγλικά δεν έχουν διαφορά. Και κατόπιν μιλήσατε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ζάμπια για να πληρωθεί την πλήρη τιμή του χαλκού. Σχετίζεται αυτό με την φορολογική πολιτική κάποιας χώρας, γιατί προξενεί εντύπωση η φορολογική πολιτική να εμποδίζει μια χώρα να πωλήσει πρώτες ύλες στην τιμή αγοράς. Μπορείτε λίγο να μας εξηγήσετε. Ναι. Και εγώ θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις για τη Ζάμπια για να καταλάβω τι συμβαίνει. Το δεύτερο θέμα. Όταν είχα πάει στην Άντις, είχαμε μια συζήτηση για την Επιτροπή Τάξ και ποιος θα είναι εκεί πέρα και πραγματικά σχεδόν ε, απέτυχε η συμφωνία. Θέλω να παίξω λίγο ένα προκλητικό ρόλο Δηλαδή, αν στείλουμε χρόνια μια διακυβερνητική επιτροπή για την φορολογία, γιατί θεωρείτε ότι θα είναι πιο αποτελεσματική από τον ΟΣΑ. Γιατί στον ΟΗΕ θα έχει πολλά μέλη, κάποιοι από αυτούς δεν θα θέλουν να λυθεί το ζήτημα, γιατί ωφελούνται από αυτές τις ροές. Μήπως υπάρχει ο κίνδυνος δηλαδή να ασχολούμαστε με τις δομές και να χάνουμε την ουσία. ότι τα λεφτά θα φεύγουν από τι αναψώμενες χώρε αν μπορούν να πάνε σε ασφαλεί χώρε όπου μπορεί ο κόσμο να κερδίσει. Ε, και πάει σε ακίνητα του Λονδίνου και σε τέτοια μέρη. Δεν πάει σε άλλες αναψώμενες χώρες, γιατί δεν έχει και νόημα. Οπότε πρέπει να κοιτάμε τι δομέ ή τι να κοιτάμε το ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο. Σας ευχαριστώ. Στρέφομαι τώρα λοιπόν στους ομιλητές μας. Δύο λεπτά ο καθένας. Ναι, ναι, θα μιλήσω και εγώ την μητρική μου, τα γαλλικά. Η κυρία Σάντον, ναι. Ναι, σα πω για την αυτόνομη την πληροφορία και όσον αφορά αυτό το report, την έκθεση αναχώρα. Πρώτα πρώτα νομίζω ότι όλε οι χώρε, οι αναπτυσσόμενε, έχουν πρόβλημα δυνατοτήτων Άρα το έχουν και οι ανεπτυγμένε χώρε όπω η Γαλλία, όσον αφορά δηλαδή το ότι υπάρχουν λιγότεροι ανθρώπινοι πόροι όσον αφορά την διαχείριση των φορολογικών θεμάτων. Άρα γι' αυτό και λέμε ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια ε, αλλά και η των πληροφοριών και οπότε κατά αυτόν τον τρόπο να υπάρχει αποτροπή όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Άρα, αποτρεπτική ε, ισχύς και επίσης να υπάρχει δυνατότητα της κοινωνίας των ε, πολιτών σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες να μπορούν να καταστήσουν ε, υπεύθυνη την ελίτ της κοινωνίας ε, κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται και σε βορρά και σε ενοδο. Για αυτό και χρειάζεται το reporting. Προχωρούμε πάρα πολύ γρήγορα βέβαια, έχουμε πολύ γρήγορες αριθμούς, αλλά παρόλα αυτά ήθελα να σας πω επ' αυτού ότι αυτό το reporting θα πρέπει να συνδέεται με την blacklist σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν πρώτα-πρώτα γιατί πρόκειται για πολύ διπλωματική διαδικασία και η λίστα δεν έχει όλες τις πληροφορίες χρειάζεται να υπάρχει πραγματικό reporting για κάθε χώρα για κάθε χώρα που γίνονται τέτοιες ε, κινήσεις. Την έχουμε αυτού του είδους ε, τις ε, δημόσιες εκθέσεις, αυτό το ε, reporting το οποίο είναι το βασικό αποτρεπτικό εργαλείο σε σχέση με την προσφυγή σε φορολογικούς παραδείσους. Άλλο πράγμα η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Κύριε Μόντες, για το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να απαντήσω στα ερωτήματα που απευθύνθηκαν απευθεία σε μένα. Κοιτάξτε τώρα, όταν είπα παράτυπος, ε, το είπα σκεμμένα. Γιατί ήταν ένα δίκτυο που ξεκίνησε μικρό και μεγά, γιγαντώθηκε πριν από 4-5 χρόνια. Προσπαθούμε δηλαδή να επισημάνουμε ότι υπάρχουν πολλές πρακτικές που σχετίζονται με την φοροαποφυγή που είναι απολύτως νόμιμες. Ένα παράδειγμα είναι η δυνατότητα και εδώ πέρα βεβαίως είναι το θέμα με τον ΩΣΑ, γιατί ο ΩΣΑ επιμένει στην αρχή της χωριστής οντότητας, δηλαδή οι χωριστές οντότητες θα πρέπει να επικοινωνούν. Οπότε είναι μετά θέμα της ε, φορολογικής αρχής να δουν τι σχέση έχουν μεταξύ τους δύο οντότητες και αν οι τιμές με τις οποίες συναλλάσσονται είναι οι τιμές αγοράς. Και όταν διαπιστώνει κάτι τέτοιο η φορολογική αρχή ότι δεν είναι η τη η τη αγορας υπαρχει αρχή της ε, απόστασης ε, δηλαδή σαν να είναι τελείως ανεξάρτητη η θηγατρική στη Ζάμπια από τη μητρική στην Ελβετία αλλά όπως είπα αν δεν μπορεί η φορολογική αρχή να αποδείξει στις αρχές της Ζάμπια πως ε, πουλάει σε χαμηλότερη τιμή ε, το χαλκό στην ελβετική εταιρεία, τότε είναι φορολογικό το ζήτημα, γιατί και οι δύο εταιρείε ε, είναι ένας όμιλος. Αλλά έτσι καταφέρουν να μειώσουν τους φόρους τους στη Ζάμπια. Ένας καθόλου νόμιμος τρόπος. Εύκολα αποδεικνύονται αυτά. Λοιπόν, τώρα για το θέμα της ε, Φορολογικής Επιτροπής. Κοιτάξτε, πριν φύγω από τον ΟΗΕ, ήμουν γραμματέας της Φορολογικής Επιτροπής του ΟΗΕ. Έχει και ο ΟΗΕ μια τέτοια. Έχει ένα δικό του μοντέλο, το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από το νοσα. Όχι τελείως διαφορετικό, τέλος πάντων έχει μια άλλη φιλοσοφία και τα μισά μέλη στην Επιτροπή ορίζονται από τις χώρες του ΟΣΑ. Γίνεται σε μια αίθουσα σαν και αυτή είναι εδώ πέρα η συνεδρίαση. Τα μέλη του ΟΣΑ είναι η μισή Επιτροπή. Οπότε ε, μιλάμε για πολύ έμπειρους ανθρώπους. Το θέμα είναι λοιπόν εάν μπορεί να χαράξει η Επιτροπή γιατί μόνο στο επίπεδο του ΩΣΑ λαμβάνονται διακυβερνητικέ αποφάσεις, γιατί η Επιτροπή του ΟΗΕ είναι Επιτροπή Ειδικών, που μόνο συστάσεις κάνει. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα για το οποίο είπαν οι αναψώμενες χώρες, Αν είναι θέμα του να θέσουμε την ατζέντα, π.χ. στον ΠΕΠΣ έχουμε αγνοήσει τελείω τις εξορρυκτικές βιομηχανίες, γιατί δεν έχουμε πρόσβαση στον Όσα; θα πρέπει να αναβαθμίσουμε την ε, Επιτροπή του ΟΗΕ. Επίσης, χρειάστηκε ο ΩΣΑ 15 χρόνια για τις κατευθυντήριες γραμμές με τις χώρες του Όσα. για να καταλήξουν σε κάποιες ε, κοινέ προδιαγραφές. Οπότε με ακόμη περισσότερες χώρες. Δεν νομίζω να γίνει γρήγορότερη η διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε για την διαφορά μεταξύ των δύο λέξεων, παράνομος και παράτυπος, και την περίπτωση της Ζαμπίας. Καλύτερα είναι να μας τα στείλετε γραπτός για να αντιληφθούμε καλύτερα το τι συμβαίνει, γιατί δεν είναι τόσο σαφές. Κυρία Σας ευχαριστώ. Όσον αφορά τι τεχνικές δυνατότητε και την αμοιβή ανταλλαγή πληροφοριών, δεν υπάρχει παντού ελευθερία στην πληροφόρηση σε πολλέ χώρε. Μόνο 19 χώρες στην ε, Αφρική έχουν τη σχετική νομοθεσία για ελευθερία τη πληροφορία και πληροφόρηση, ε, αλλά δεν υπάρχουν και συγκεκριμένε ε, διατάξει για την ανταλλαγή των φορολογικών. Άρα το θέμα είναι η δουλειά του κόσμου. Όλα αυτά σημαντικά για την διακυβέρνηση. Να έχει δηλαδή ο κόσμος προσβασιμότητα, αλλά και να λειτουργεί για το σύστημα ε, εύρυθμα. Καλύτερη διαφάνεια, να υπάρχουν κάποια μητρώα για τις εταιρείε και έκανα έρευνα πριν πέντε χρόνια και κοίταξα αυτό το μητρό των εταιριών να δω τι μπορώ να βρω και είχαμε ε, δεν είχαμε καμία επικαιροποίηση, ιδίω όσον αφορά τις πολυεθνικές. Υπάρχουν επομένω κάποια δημόσια μητρώα, αλλά τα μητρώα αυτά δεν ενημερώνονται. Κάτι άλλο τώρα, κάτι το οποίο νομίζω έχει να κάνει και με την ε, Ζάμπια. Αυτές οι μυστικές συμβάσεις, τα συμβόλαια μεταξύ κυβερνήσεων και εταιριών. Αυτό είναι μια μαύρη τρύπα. Κανείς δεν μπορεί να τα δει αυτά. Άρα υπάρχει η κερδοσκοπία, είναι προβληματικό. Άρα ούτε εδώ υπάρχουν πληροφορίε τώρα όσον αφορά την ε, Φορολογική Επιτροπή ήταν πολύ σημαντικό αυτό που έγινε και πριν από δύο χρόνια είχαμε μια μελέτη που έλεγε για τη διπλή φορολογία ε, στα πλαίσια του ΟΣΑ, μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ και μεταξύ χωρών ΟΣΑ και τρίτων. Και όταν ε, υπήρχαν τέτοιες συμφωνίες χρησιμοποιούσαν το πρότυπο του ΟΗΕ μεταξύ τους. Με τρίτες χώρες όμως χρησιμοποιούσαν το δικό τους μοντέλο του ΟΣΑ. Και από ό,τι κατάλαβα οι χώρες του ΟΣΑ έχουν ένα πρότυπο, ένα στάνταρ καλό για αυτές, γιατί είναι στο ίδιο επίπεδο ανάπτυξης. Οπότε τα βρίσκουν ε, όταν κάνουν συμβάσει με την άλλη. Όταν όμως έρχεται η ώρα επαφής με τρίτη χώρα, ε, τότε ε, η, ισορροπία των δυνάμεων είναι υπέρ των χωρών του ΩΣΑ. Οπότε το ρυθμίζουν έτσι και έτσι δεν υπάρχει ένα δημοκρατικό έλλειμμα. Γιατί δεν υπάρχει ισότητα για τις σχετικές επαφές. Άρα, για κοιτάξτε τι γίνεται στις διακοινοβουλευτικές διασκέψεις. Τι γίνεται με τις χώρες που δεν έχουν κληθεί, που δεν συμμετέχουν. Αν κάνετε τη σύγκριση, τον παρελισμό θα καταλάβετε. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα ολοκληρώνουμε αυτή την ε, συζήτηση, δίνοντας το λόγο στον κύριο Κόφο, τον εισηγητή μας. Ευχαριστώ το πάνελ πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι πληροφορίες και η συζήτηση. Μα καν είχαμε χρόνο για να καλύψουμε όλα αυτά τα οποία είπατε. Έχουμε πολλά αξιόλογα τα οποία αναφέρθηκαν και τα κρατάμε για την δική μας δουλειά εδώ, στην Επιτροπή μας. Για ό,τι κάνετε επομένως είμαι ευγνώμονας. Να μην ξεχνούμε ότι έχουμε τεράστια ευθύνη να έχουμε συνέπεια στις πολιτικές μας. Όταν επομένως νομοθετούμε για τα φορολογικά εδώ και φτιάχνουμε πολιτικές φορολογικές, θα πρέπει να σκεφτόμαστε τις αντισώμενες χώρες. Άρα, πολύ σημαντική συνέπεια. Και όπως ε, είπατε στην αρχή, σε εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να χορηγείται αναπτυξιακή βοήθεια από τη μία και από την άλλη όμως έχουμε μεταξύ μας κάποια διαρθωτικά προβλήματα όσον αφορά την οροφή που διέπει τα έσοδα για τις τρίτες χώρες. Και είπαμε ότι είναι αδίκημα η φοροδιαφυγή. Αυτό πρέπει να το λύσουν οι αντισώμενες χώρες. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, πιο σημαντικό από την αναπτυξιακή βοήθεια. Τώρα για τα θέματα που αναφέρατε ειδικότερα. Αρχίζω από το τέλος. Μίλησατε για τη σχέση των πλαισίων ΟΣΑ και ΟΗΕ για σύμφωνες διπλής φορολόγησης. Μα αν υπάρχει ανισορροπία δυνάμεων, τότε παραβαίνουμε την αρχή μας της ε, δίκαιης συνεργασίας, συνεργασίας υπό ίσους όρους. Άρα υπάρχει πρόβλημα και θα πρέπει να επιληθεί. Τώρα όσον αφορά ε, αυτό το σύστημα των εκθέσεων αναγόρα. τον ίδιο το πόσο σημαντικό είναι. και για τη σχέση με τις όμορες χώρες. Τα έχουμε πει εδώ, τα έχουμε πει και αλλού. Και έτσι θα μπορέσουν οι χώρες να εξασφαλίσουν το ότι οι εταιρείε θα πληρώνουν τους φόρους. Πας μια εβδομάδα ήρθαμε σε επαφή με την Παγκόσμια Τράπεζα Υπάρχουν προγράμματα εισπραξής των φόρων και δαπανών από πλευράς κρατικής. Ρίχνει μια ματιά και στα Panama Papers. Εδώ έχουμε δύο τινά. Πρώτα-πρώτα τις δυνατότητες της ε, κυβέρνησης να ε, φορολογεί δίκαιο και από άλλη μεριά όμως έχουμε αυτά τα οποία αναδύθηκαν σαν προβλήματα. Τα σκάνδαλα που οδήγησαν και στην παρέτηση του Πρωθυπουργού της Ισλανδία, για παράδειγμα. Μα αυτά υπάρχουν και στις αντισώμενες χώρες. Οπότε βλέπουμε ότι πολλέ φορέ υπάρχει πολιτική αντίσταση για περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη ενέργεια πληροφοριών. Γιατί έτσι προστατεύεται η πολιτική ελίτ. Άρα και αυτό θα πρέπει να το επισημάνω. Τώρα, για τις μαύρες λίστες, πρόεδρε. Θα πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη εδώ. Να προβλέπονται κάποιες κυρώσεις για όσους δεν συνεργάζονται. Περί αυτού πρόκειται εδώ. Απαρίθμηση των φορολογικών παραδείσων. Των μη συνεργαζομένων. Μπα και έτσι τους πείσουμε να είναι πιο συνεργάσιμοι. Τώρα για τον όσα... Σαν αφορά τώρα το BEPS, εγκρίθηκε από το G20. Βοήθεια προς τις χώρες αλλά εκτός από τις πολύ πλούσιες χώρες ε, πολλές φορές και οι λιγότερο πλούσιες θέλουν να προστατεύσουν τα συμφέροντα των λιγότερων επιτυγμένων χωρών. Άρα τέλος πάντων θα πρέπει στα πλαίσια του ΟΣΕ να εξασφαλίσουμε την συμμετοχή των λιγότερων επιτυγμένων χωρών έτσι θα λυθούν πολλά προβλήματα. Νομίζω μακρηγόρησα, Πρόεδρε, αλλά ήταν πολλά τα αξιόλογα που άκουσα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοφότ. Και ευχαριστώ και όλους τους προσκεκλημένους για τις πληροφορίες τους. Στρέφομαι τώρα στα μέλη της Επιτροπής ΔΕΒΕ. Θέλω να σας πω ότι αποφασίσαμε για το σχέδιο έκθεσης του Γεπε και του Μικαήλ Τόιερ που τώρα υπάρχει σε όλες τις γλώσσες, την προθεσμία τη θέσαμε στην 31η Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Οπότε, αν υπάρχουν τροπολογίες που ενδιαφέρουν την δικιά σας Επιτροπή, ευχαρίστως να τις λάβουμε υπόψη μας. Τώρα, Λίντα, εσύ για το δεύτερο πάνελ. Ευχαριστώ πολύ θίξαμε πολλά ζητήματα που θα επανέλθουν σίγουρα στο δεύτερο πάνελ που έχει να κάνει με το ρόλο των αναπτυσσόμενων χωρών στη δημιουργία ενός διεθνούς φορολογικού συστήματος. Τρεις ομιλητές έχουμε. Τον κύριο Σάβιορ Μουάμβα από την Action Aid στη Ζάμπια, οπότε θα μας βοηθήσει. Στη συνέχεια έχουμε τον Tove Riding από τη Eurodad, για την φορολογική δικαιοσύνη και τον κύριο Σολ Πιτσότο που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ. Αρχίζουμε λοιπόν με τον κύριο Σάβιο Παμπουά και ίσως μπορείτε να μας διευκρινίσετε τα περί Ζάμπια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Όντω δουλεύω για την Action Aid International αλλά και για την Ζάμπια. Έχω δουλέψει στη Ζάμπια λοιπόν για μια υπόθεση μετά από προσφυγή στον ΟΣΑ όσον αφορά διεθνείς επιχειρήσεις κατά της Γκλέγκο από διάφορες ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις στο ελβετικό σημείο επαφής. Εκεί ακούστηκαν βέβαια διάφορα πράγματα σαν και αυτά που ακούσαμε και εδώ. Ξεκινήσαμε από έναν έλεγχο που έγινε από τις αρμόδιες αρχές στην Ζάμπια που έδειξε ότι η Γκρέγκο χρησιμοποιούσε διαφορετικούς τρόπους στις, συνολ... στις συναλλαγές και μείωνε τους φόρους που έπρεπε να πληρώσει στη Ζάμπια είτε με πωλήσει χωρίς αποδεικτικά στοιχεία μέσω των θυγατρικών και ήταν πολύ δύσκολο να αποδεχτεί σε τι τιμή έγιναν οι πωλήσει. Το θέμα είναι ότι έπρεπε να αναθεωρηθούν οι χρώσει της εταιρεία απέναντι στην ε, Ζάμπια μετά από την έκθεση αυτή. Έγιναν πληρωμές ε, στον ε, Μαυρίκιο, ενώ δεν είχε καθόλου δραστηριότητες εκεί. Όλα αυτά συνδυαζόμενα κατέληξαν στο ότι Γκλένκο πράγματι εφάρμοζε μια επιθετική φορολογική τακτική και έδινε και λάθος λογιστικά βιβλία. Αυτό είναι το πρόβλημα όμως τώρα, γιατί πότε πρόκειται για φοροδιαφυγή και πότε για φοροαποφυγή. Τι είναι παράνομο και τι όχι. Είναι δύσκολο να πει κανείς με σιγουριά κατά πόσο οι πρακτικές αυτές των επιχειρήσεων είναι παράνομες ή όχι. Δεν θα σταθώ περισσότερο σε αυτό. Πάντως, 50 εκατομμύρια δολάρια φαίνεται ότι σε δύο χρόνια έχασε η Ζάμπια από την μία αυτή επιχείρηση. Χρήματα τα οποία έδωσε στη Ζάμπια το Ηνωμένο Βασίλειο για στήριξη. Καταλαβαίνετε λοιπόν την έλλειψη συνοχής. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να, να δίνει χρήματα στη Ζάμπια για να την βοηθήσει, όταν η Ζάμπια χάνει χρήματα από ευρωπαϊκέ πολυεθνικέ. Για σκέψη όλα αυτά. Τώρα, θέλω να φερθώ σε δύο ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή σας για την έκθεση αυτή και για την πρόσκλησή σα να έρθουμε και να σχολιάσουμε. Είναι πολύ σημαντικό και θετικό που τίθεται εδώ η σχέση με τα διεθνή ζητήματα και για τους εθνικούς παράγοντες που οδηγούν στην φοροαποφυγή. Η σχέση μεταξύ του τι συμβαίνει στην Ευρώπη και τις επιπτώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι κάτι που δεν υπογραμμίζεται επαρκώς την έκθεση κατά τη γνώμη μας. Πρέπει να αναφερθούμε σε συγκεκριμένα φορολογικά μέτρα τα οποία πήραν ή δεν πήραν οι ευρωπαϊκές χώρες για τη διαδικασία PEPS τη διαδικασία, έτσι. Είναι σαφές ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν έχουν συμμετάσχει επαρκώς μέχρι τώρα. Και όπως είπε και κάποιος, το αποτέλεσμα είναι ότι το ΠΕΠΣ e υπογραμμίζει πράγματα που αφορούν πιο πολύ τις αναπτυγμένες χώρες. Φορολογικές συμφωνίες, συνθήκες, η εξοριστική βιομηχανία είναι πράγματα στα οποία δεν έχει δοθεί επαρκής προσοχή. Η Αφρικανική όμως έκθεση τι λέει. Λέει ότι τα περισσότερα προβλήματα είναι με τον εξορρυκτικό τομέα. Στις χώρες δηλαδή Νιγηρία, Μοζαμβίκη, Αγκόλα, Νότια Αφρική, Ζάμπια, χώρες δηλαδή που έχουν μεγάλη εξορρυκτική βιομηχανία, εκεί υπάρχει η μεγαλύτερη απώλεια χρημάτων. Πρέπει λοιπόν, αν υπήρχε μάλλον αρκετός χρόνος για τη συμμετοχή και των χωρών αυτών, ίσως το BEPS έχει καταλήξει κάπως διαφορετικά. Τώρα προτείνεται η υποανάπτυξη χώρες να εφαρμόσουν αυτό το οποίο έχει συμφωνηθεί. Μα δεν μπορείτε να καλέσετε ποδοσφαιριστές να παίξουν σε έναν αγώνα του οποίου τους κανόνες έχουν αποφασίσει κάποιοι άλλοι στα κρυφά. Πρέπει να ανοίξει λοιπόν ο χώρος. Να υπάρχει ένα διακυβερνητικό σώμα στη ΛΟΙΕ. Η δημοκρατία κοστίζει. Έχει κάποιο τίμημα. Μερικές φορές πρέπει να επιβραδύνουμε, να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο χρόνο αν θέλουμε να καταλήξουμε σε κάτι που να έχει νόημα. Μπορεί να υπάρχουν τα προβλήματα που γνωρίζουμε στο σύστημα του ΟΗΕ, αλλά ίσως να αξίζει το κόπο. Τέλος, για τις ε, συνθήκες, συμφωνίες φορολογικές, είτε πρόκειται για την Κλένκο, είτε πρόκειται για την, στη Ζάμπια, είτε για την Ουγκάντα, όπου και εκεί 200 εκατομμύρια περίπου δεν πλήρωσε μια εταιρεία. Απλώς και μόνο επειδή μεταφέρθηκε το Μαυρίκιο, επειδή υπάρχει συμφωνία Ουγγάντα-Μαυρίκιος. Ε, Τεράστιες απώλειες. Έχει μεγάλη σημασία να αντιμετωπίσουμε αυτά τα αρνητικά ζητήματα και να δούμε τα φορολογικά δικαιώματα πώς ε, και πού ισχύουν. Έχουμε εδώ την έκθεση και online μπορείτε να τη βρείτε όπου αναλύουμε 500 συμφωνίες ανάμεσα σε αναπτυσσόμενες χώρες και ευρωπαϊκές χώρες. Και τις ταξινομήσαμε από το ποιες είναι οι πιο περιοριστικές συμφωνίες στις λιγότερο περιοριστικές. Ποιες ευρωπαϊκές χώρες λοιπόν υπογράφουν τέτοιες συμφωνίες. Έτσι θα δείτε και τις δικές σας χώρες. Το Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα είναι ένα από αυτά που έχει πολύ περιοριστικές ε, συμφωνίες. Πολιτική συνοχή, συνοχή στις εμπορικέ πολιτικές. Και αυτές οι συμφωνίες εμπορικέ εμπορικές επηρεάζουν την συλλογή φόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η διαδικασία ΠΕΠΣ λοιπόν, σας είπα, ελεκτικά ζητήματα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ κυρία Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω από ένα σωστό ερώτημα που αναφέρατε πριν. Δηλαδή, αν προσκαλούμε τις αναψώμενες χώρες όταν συζητάμε αυτούς τους κανόνες μήπως θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί μια συμφωνία. Ναι, ε, έτσι είναι η δημοκρατία. Και νομίζω πως εμείς ε, στην Ευρώπη συνήθως ακολουθούμε αυτές τις αρχές και ειδικά για φορολογικά ζητήματα δεν αντιλαμβάνουμε πως η Ευρώπη υπερασπίζεται ένα σύστημα στο οποίο πάνω από 100 χώρες αποκλείονται και εκεί πέρα καθορίζονται οι κανόνες. Και ναι, πρέπει να εφαρμοστούν στις χώρες που δεν ήταν παρούσες και για τις οποίες δεν είναι νομικά δεσμευτικές. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη πίεση στις αναψώμενες χώρες παρά το ότι δεν είναι δεσμευτικοί αυτοί οι κανόνες για αυτές. Μια απόφαση που έχει λάβει ο ΣΑ από πολλά χρόνια είναι πως εάν μια εταιρεία λειτουργεί σε δύο χώρες τότε το δικαίωμα φορολογίας ε, της εταιρείας θα πρέπει να είναι κατά κύριο λόγο στην ε, χώρα όπου είναι η έδρα της εταιρεία αυτό, παρά το ότι όλο και περισσότερες χώρες έχουν πλέον έδρα εταιριών, ε, κατά κύριο λόγο οι έδρες είναι στις χώρες του ΟΣΑ. Και αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν θέλουν να δεχτούν τους κανόνες του ΩΣΑ γιατί ο ΩΣΑ έχει αποφασίσει κανόνες που τον ωφελούν. Το άλλο παράδειγμα του γιατί διστάζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι αυτή η αρχή της απόστασης η λεγόμενη που δεν λειτουργεί στις αναπτυσσόμενες χώρες και μάλιστα ούτε οι χώρες του ΩΣΑ δεν έχουν καταφέρει να την κάνουν να λειτουργήσει. Τώρα δεν θα κατηγορήσω κανένα σας αν δεν έχει διαβάσει τα αποτελέσματα του BEPS γιατί είναι 1900 σελίδες. Αν προσπαθήσετε όμως ένα ζήτημα που θα σας ε, καταπληξεί είναι το πόσο λίγο έχει αλλάξει αυτή η αρχή της απόστασης. Επίσης, στον κατάλογο των επίμαχων αποφάσεων του ΩΣΑ θα προκύψουν και άλλες μετά τον ΠΕΠΣ. Ένα από τα πράγματα τα οποία αποφάσισε είναι πως οι, χώρες, οι αναφορές αναχώρα πρέπει να είναι μυστικές. Και αυτό μάλιστα αντιβαίνει σε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έλεγε πως θα έπρεπε να είναι δημόσιε. Ευτυχώ η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωράει πια πέρα από τον ΠΕΠΣ όπως και πολλές άλλες χώρες. Επίσης αναφέρθηκαν τα patent box. Θα δείτε τώρα στον ΠΕΒΣ πω υπάρχει μια περιγραφή του πώ πρέπει να γίνονται αυτά. Θα είναι μια νέα επιβλαβή ε, φορολογική πρακτική και έχουμε χώρες όπως η Ιρλανδία που λένε εγώ εφαρμόζω την BEPS ε και άρα θα φέρω ένα patent box. Πριν αρχίσουμε λοιπόν να μιλάμε για το αν είμαστε υπέρ ή κατά, θα πρέπει να δούμε το τι είναι το BEPS. και βεβαίως ε, θα ε, ζητήσουμε και θα, θα έχουμε και περισσότερες αποφάσεις με τρόπο αντιδημοκρατικό. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχει κάνει συχνά όσα είναι να μαζεύονται κάποιες χώρες ε, G20 και να υιοθετούν κανόνες. Και μετά μόλις εγκριθούν αυτοί οι κανόνες λέμε ωραία ακολουθήστε τις και οι υπόλοιποι. Αυτό έγινε πρώτη φορά στην ανταλλαγή πληροφοριών, όπου ενέκριναν τους κανόνες και μετά υπήρχε το λεγόμενο Παγκόσμιο Φόρουμ, όπου μπορούσαν οι υπόλοιπε χώρε να έρθουν και απλά να ακολουθήσουν. Τώρα έγινε ακριβώς πάλι το ίδιο με τον ΠΕΠΣ. Τους λέγαμε δύο χρόνια πρέπει να μπουν και οι άλλες χώρες στην ΕΦΣΑ. Μόλι εγκρίθηκαν οι κανόνε, ε, προσεκλήθησαν οι άλλε χώρε εάν ήθελαν να συμμετάσχουν στην εφαρμογή. Και μόλις υπογράψουν βεβαίως τις 1900 σελίδες τις συγκεκριμένες, αν υπάρχουν κενά και υπάρχουν κενά, μπορούν να συζητήσουν το πώς θα καλυφθούν αυτά τα κενά. Αλλά αυτό είναι μεγάλη δέσμευση για μια αναπτυσσόμενη χώρα που δεν ήταν στις διαπραγματεύσεις. Τώρα για το τελευταίο ερώτημα αν του προσκαλέσουμε όλους μήπως θα ε, γεμίσουμε φορολογικούς παραδείσου. Δηλαδή εκπλήσωμε ότι μετά τα Lux Leaks και τα Swiss Leaks και το τι συμβαίνει στην Ολλανδία ακούμε αυτά τα επιχειρήματα ότι οι αναπτυσσόμενε χώρες είναι φορολογική παράδειση. Η φορολογική παράδοση δεν είναι ότι αν ξεφορτωθούμε κάποιους ε, τουλάχιστον έχουμε κάνει κάποια πρόοδο και μια μαύρη λίστα που θα περιλαμβάνει μόνο λίγες χώρες δεν λειτουργεί. Γιατί, γιατί είναι φορολογικός ανταγωνισμός. Προσφέρουν ένα προϊόν σε ανθρώπους που θέλουν να αποφύγουν φόρους. Και τι θα κάνουμε, αν βάλουμε κάποιες χώρες στη μαύρη λίστα και όχι όλες, είναι ότι θα βοηθήσουμε την Ελβετία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία και τις ΙΠΑ αυτού του πλανήτη. Θα τις βοηθήσουμε στον ανταγωνισμό, γιατί να έχετε κατά νου πως υπάρχουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες και οι που δεν ανταλλάσσουν πληροφορίες αυτομάτως αυτή τη στιγμή με αναπτυσσόμενες χώρες και δεν δεσμεύονται για να ακολουθήσουν τους κανόνες του ΩΣΑ. Αυτό είναι λοιπόν ο φορολογικός ανταγωνισμός. Είτε τα αντιμετωπίζουμε όλες τις χώρε, είτε δεν κάνουμε τίποτα. Θα πηγαίνουν τα λεφτά από τη μια χώρα στην άλλη. Τέλος. Δεν πρέπει να έχουμε ένα φορέα του ΟΗΕ για να είμαστε ευγενικοί με τι αναψώμενες χώρες. Πρέπει να το κάνουμε και για εμάς. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα παγκόσμιο σύστημα. Υπάρχουν πάνω από 100 χώρες που δεν ήταν στην αίθουσα όταν αναπτύχθηκε αυτό το σύστημα και δεν έχουν καμία υποχρέωση να τα ακολουθήσουν. Χώρε όπω η Βραζιλία και η Κίνα ε, ακολουθούν δικό του δρόμο, δικού του κανόνε. Όλο και περισσότερε αναπτυσσόμενε χώρε προσπαθούν να στήσουν διαφορετικά φορολογικά συστήματα. Οπότε θα δημιουργηθεί χάο εάν ε, θέλουμε εμεί να θέσουμε του κανόνε για τι αναπτυσσόμενε χώρε. Και αυτό μετά θα δημιουργήσει περισσότερα παραθυράκια, περισσότερη φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή και περισσότερο χάο. Και θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου το σύστημα θα είναι τόσο περίπλοκο ώστε την επόμενη φορά θα είναι δίπλα μου πολυεθνικές και θα ζητάνε μια πραγματική παγκόσμια διαπραγμάτευση. Ε, οδεύουμε προς χάος. Δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα. Όχι και πολύ αισιόδοξα αυτά. Περνάμε τώρα στον επόμενο μιλητή. Ο καθηγητής Σόλ Πιτσότο. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Έστειλα ένα έγγραφο για την παρουσίασή μου, αλλά επειδή δεν έχουμε χρόνο, εγώ τώρα θα σας δείξω κάποια συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένα το ζήτημα της τιμολογικής πολιτικής, της διαμόρφωσης των τιμών δηλαδή ε, και ασχολούμαι με το Διεθνές Κέντρο για ε, Φορολογική Πολιτική και Ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο και κάνουμε έρευνα για διάφορους ε, φόρους αλλά κυρίως για τους διεθνείς φόρους και επίσης είναι σαφές ότι αν οι πιο μεγάλες εταιρείε στον κόσμο μπορούν να εκμεταλλευτούν τα φορολογικά συστήματα για να πληρώσουν περισσότερο φόρο. Αυτό έχει επιπτώσεις στην ε, φορολογία όλων. Επίσης ασχολούμαι και με το δίκτυο BEPS που έχει διεθνή χαρακτήρα και ασχολούμαι με όλα τα BEPS από ε, ε, τη διάβρωση βάσης και, τα, και κέρδη και βλέπουμε επομένως ότι υπάρχουν πολλά θέματα εδώ και η εντολή για το Project BEPS προήλθε από το G20 ούτως ώστε να μεταρρυθμιστεί το δίκαιο ούτως ώστε ε, να φορολογηθούν εκεί που ασκούν δραστηριότητα οι πολυεθνικές. Αλλά βέβαια θα πρέπει κάθε χώρα να είναι κυρίαρχη να θεσπίσει τους νόμους που θέλει. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση γιατί είναι σαφές ότι αν δεν υπάρχει συντονισμός στην νομοθεσία ε, τότε ε, μάλλον είναι ε, ε, φαντασίωση το είναι να ε, φορολογήσουμε τις πολυεθνικές. Οπότε όλα αυτά μας απασχολούν στο Project BEPS και έχουμε δημοσιεύσει στο ICDD διάφορα από αυτού και κυρίως ασχολούμαστε με το transfer pricing την τιμή μεταβίβαση, τιμολόγηση, τι είναι. Τέλος πάντων έχουμε διάφορες εκθάσεις ε, που αφορούν το project BEPS και έχουμε να θεωρήσει τις καθεντήρες για το transfer pricing και ακόμα όμως έχουμε πολλά να κάνουμε κυρίως όσον αφορά την ε, μέθοδο <clears throat> της παράκαψης νομοθεσίας για τα κέρδη και προσπαθούμε επίσης να δούμε τι γίνεται με την φορολογία που επιβάλλεται στην ε, πηγή, αλλά θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Θα πρέπει να δούμε σε λεπτομέρεια ε, και κάποια τα οποία είπαν ε, προλαλήσαν τα δούμε είναι σωστά ε, γιατί οι βασικές χώρες του ΩΣΑ συνήθως είναι εξαγωγικές χώρες αλλά κάποιες άλλες είναι εισαγωγικές και φυσικά οι πολυεθνικές κάνουν εισαγωγές και εξαγωγές οι αναπτυσσόμενες χώρες συνήθως δεν έχουν δικές τους πολυεθνικές έχουν κάποιες χώρες τώρα που είναι στο G20 άρα το BEPS έχει ωφελήσει τώρα ε, κάποιες ε, χώρες που είναι εξαγωγική η οικονομία τους. Και γι' αυτό και έχουμε και αυτές τις ε, καθεντήρες γραμμές για το transfer pricing. Σε γενικέ γραμμές, ό,τι αλλαγές έχουν γίνει μέχρι τώρα στις καθεντήριες γίνονται ούτω ώστε να έχουμε καλύτερη προσέγγιση. Δηλαδή, να έχουμε μια λειτουργική ανάλυση, να εξετάζουμε την πολυεθνική, όχι σαν μια ε, μονάδα, να θεωρούμε ότι είναι μια εταιρεία πολυεθνική, αλλά όπως ε, ε, ήδη αναφέρθηκε να έχουμε την ισχύ των κανόνων του όσα Λέει ο ΩΣΑ πρέπει να εξετάζουμε την κάθε πολυεθνική χωριστά σε κάθε χώρα. Όμως θα πρέπει να τις εξετάζουμε σύμφωνα με τη λειτουργία τους και έτσι να ξέρουμε στο τι μοντέλο επιχειρησιακό έχει κάθε πολυεθνική και να δούμε μετά τι λειτουργίες ε, υπάρχουν και τι γίνονται τα κέρδη ανάλογα με τις βασικότερες λειτουργίες τους. Άρα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα άλλα περιουσιακά στοιχεία, τι γίνεται με το κίνδυνο και άρα εξετάζεται η λειτουργία που αφορά στον έλεγχο αυτών των μεταβλητών. Άρα όπου υπάρχει σημαντική δραστηριότητα πολυεθνικής και έχει και κάποια συνεργαζόμενη εταιρεία, εάν εκεί δεν ασκείται ο έλεγχος, τότε αυτή η συνεργαζόμενη εταιρεία έχει αυτά που ονομάζουμε καθημερινά μπανάλ ε, έσοδα. Ας πούμε το Google στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν ξέρουν τις λεπτομέρειες, απετέλεσε στόχο των ε, φορολογικών αρχών. Οι δραστηριότητες εκεί ε, θεωρείται ότι παρά το ότι έχει χίλιους μηχανικούς στη χώρα και 3.000 ανθρώπους που ασχολούνται με το μάρκετινγκ, θεωρούμε ότι πρόκειται για συνήθεια δραστηριότητα, καθημερινή κοινή δραστηριότητα. Ε, αν ο έλεγχος γίνεται από το εξωτερικό, τότε έχουμε κάποιες ε, ε, αντίστοιχα βρετανικές πολυεθνικές που ε, ελέγχουν εταιρείε που βρίσκονται σε άλλη χώρα. Άρα τα κέρδη έρχονται στον Ηνωμένο Βασίλειο. Να, γιατί είναι λάθος το μοντέλο του όσα το θέμα επομένω είναι το αν η δραστηριότητα είναι κοινή ή όχι, ανεξάρτητα της έκτασης που έχει. Αυτό αφορά και την έρευνα Τώρα έχουμε δραστηριότητες ερευνητικές ε, και αναπτυξιακές σε Ινδία, ε, Κίνα, Μεξικό και, και, σε άλλες χώρες έχουν και τις αναπτυξιακές δραστηριότητες από τις φαρμακευτικές εταιρείε που κάνουν τις δοκιμές στους εμπεσόμενες χώρες αλλά ε, αυτό θα το σύμφωνα με αυτές τις καθεντήριες ως λειτουργία κοινή. Για πολλούς λόγους, εδώ πέρα πάσχει αυτό το μοντέλο και ιδίως, να κοιτάξτε εδώ πέρα στο τέλος της ε, προσιάσεως μας, ότι έτσι θα πρέπει οι, οι, οι αρχές να έχουν μία προσέγγιση κατά περίπτωση ε, γιατί θα πρέπει να δούμε πώς οι χώρες μπορούν να δημιουργήσουν δυνατότητες παραγωγικές ε, αλλά δεν θεωρούμε ότι αυτή είναι βιώσιμη η προσέγγιση για το διεθνέ φορολογικό δίκαιο. Χρειάζεται το ίδιο το φορολογικό δίκαιο αναθεώρηση. Υπάρχουν εναλλακτικέ προσεγγίσεις σε κάποιες χώρες. Η Βραζιλία είχε ένα σύστημα σταθερού ε, περιθωρίου. Ε, αυτό ήταν ε, εύκολο, ήταν εύχριστο από πλευρά των φορολογικών υπαλλήλων και ούτε ήταν περίπλοκο ο ΣΑ θα πρέπει να έχει ένα ε, κουτί εργαλείων όπως ονομάζεται, εργαλειοθήκη και υπάρχει και το σύστημα του ασφαλούς λιμένα. υπάρχει η τροποποιημένη ε, μέθοδος ε, καθαρού περιθωρίου και οπότε έχουμε εδώ πέρα σαν σημείο αναφοράς το κέρδος της εργαζόμενης εταιρείας σαν ποσοστό του κέρδους της ε, ομάδας, του ομίλου, του εταιρικού. Και αυτό το χρησιμοποιεί το μοντέλο και η Αμερικανική φορολογική αρχή σε σχέση με κάποιο είδους 25% επί του τζίρου που είναι το εισόδημα, το ελάχιστο εισόδημα προεπιβολής των φόρων να τι θα μπορούσε να κάνει ο ΩΣΑ για μια πιο εύκολη λύση. Όμως μέχρι τώρα ε, το, το, το BEPS δεν έχει ασπαστεί αυτές τις θεωρίες. Έχουμε το BEPS 2 και η θεωρία split profit ε, θα έπρεπε να έχει εξεταστεί. Πάντως οι χώρες του ΩΣΑ θα προσπαθήσουν να περιορίσουν το πώς θα εξελιχθεί αυτή η μέθοδος split profit. Και να αναπτυσσόμενες τώρα εμένουν να υπάρξει μια εναλλακτική προσέγγιση. Πάντως η Επιτροπή σας θα μπορούσε να βοηθήσει ότι κάθε εκδοχή του BEPS να βοηθήσει και να υπάρξει μια πιο κατάλληλη, πιο δόκιμη προσέγγιση. Να μην γίνονται πάλι τα ίδια και τα ίδια. Και να βρεθεί μια λύση που θα ωφελήσει και μόνο τι αναπτυσσόμενε, αλλά όλε τι χώρε. Ευχαριστώ. Εμεί ευχαριστούμε πολύ ενδιαφέροντα όσα είπατε που αναδεικνύουν τα προβλήματα. Η Άννα Γκόμες έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ για όλα αυτά που ακούσαμε. Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κάθε φορά που προσπαθούμε να σχεδιάσουμε φορολογικά συστήματα. Φοβούμε όμως ότι δεν θέλουμε απλώς να σχεδιάσουμε ένα φορολογικό σύστημα απλό, με διαφάνεια, που να μην αφήνει περιθώρια για διαφθορά κλπ. Συγχρόνως έχουμε να κάνουμε και με φορολογικούς παραδείσους. Συνεπώς, έχουμε εξάγει συστήματα διαφθοράς σε ολόκληρο τον κόσμο. Κανείς δεν έχει να δώσει μαθήματα σε άλλους και όντω αυτά που έχουν αντιγράψει άλλες χώρες αποτελούν την επέκταση αυτών που κάνουμε εμείς εδώ. Χώρες όπως η δικιά μου ακούνε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για να επενδύσουμε στην υγεία, στην εκπαίδευση, σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες. Τα χρήματα όμως υπάρχουν και είναι κολλημένα σε φορολογικούς παραδείσους. Και σίγουρα αυτό συμβαίνει και σε πολλές άλλες χώρες, κυρίως σε αναπτυσσόμενες χώρες και έχουμε τεράστια ευθύνη εμείς. Υπάρχει τεράστια αντίφαση. Έχουμε μια αναπτυξιακή πολιτική που έχει σαν στόχο να βοηθήσει την ανάπτυξη ικανοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες και από την άλλη μεριά εξακολουθούμε να έχουμε ένα φοβερό σύστημα φορολογικό το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα όλων των φορολογούμενων και των πολιτών άλλων χωρών. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, διαπίστωσα την ηρωνία της κυρίας Ράιντινγκ, οπότε τελικά όντως πρέπει να καταπολωμηθεί το απόρριτο. Και ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό που, μπορεί, που προσπαθεί να πετύχει η Επιτροπή μας, τάξ. Και ίσως και στα πλαίσια της επόμενης Επιτροπής που θα φτιάξουμε για τα έγγραφα του Παναμά. Πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε και αυτό προτείνεται, να καταπολεμήσουμε το απόρριτο. Όταν ξέρουμε ότι τώρα υπάρχουν κλεπτοκρατίες και στις συναψόμενες χώρες αλλά και σε άλλες που βασικά αυτό θέλουν, να διατηρηθεί το σύστημα και το απόρριτο. Ευχαριστώ η Μαρία Γόιμπουκ. Ευχαριστώ Ευχαριστώ επίσης για τις πολλές ε, πληροφορίες και πραγματικά έχουμε μία ιδιαίτερη αντίληψη της ε, συνέχειας της πολιτικής Αν από τη μία έχουμε αυτά τα παραθυράκια αυτό που αναφέρθηκε η ηρωνία στο σύστημα που ωφελούν κάποιους ανθρώπους και τα επιμένουμε να τα διατηρούμε και από την άλλη δίνουμε γενναιόδορη αναπτυξιακή βοήθεια Δηλαδή, τι συνέπεια στην πολιτική μας είναι αυτή. Θα πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια σε όλους τους τομείς της πολιτικής και στην εμπορική πολιτική και στην αναπτυξιακή. Και να επανεξετάσουμε, όπως είπα, όλους τους τομείς. Έχουμε τους στόχους της χιλιετίας. και θα πρέπει να προσαρμοστούν όλοι οι τομείς της ε, πολιτικής. Επίσης, αυτή τη στιγμή γίνεται αυτή η συζήτηση στο πλαίσιο του G20 και του ΟΣΑ, οπότε 80% των χωρών παγκοσμίω αποκλείονται από τη συζήτηση. Πώς θα μπορούμε λοιπόν να έχουμε μια διαδικασία που θα συμπεριλαμβάνει και τις χώρες αυτές για να υπάρχει μια παγκόσμια διακυβέρνηση όπως αναφέρθηκε. πώς θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε κοινού κανόνες ε, και να έχουμε μια κοινή βάση για φορολογική πολιτική και φορολογικά ζητήματα. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι πως θα ήταν καλύτερο να απτύξουμε κοινούς κανονες και να εχουμε ένα νέο διακυβερνητικό φόρουμ για την διεθνή συνεργασία σε φορολογικά ζητήματα υπό την αιγίδα του ΟΗΕ όπου θα συζητάμε όλα αυτά τα ζητήματα με μια ευρύτατη εντολή του ΟΗΕ. Πρέπει να έχουμε λοιπόν μια βάση όπου θα μπορούμε να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα και προβλήματα. Στα τωρινά φόρα μάλλον δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Κάποιος άλλος συνάδελφος θα ήθελε τον λόγο. Άλλη μία ερώτηση προς τον καθηγητή τον κύριο Πιτσότο για τα ζητήματα που είπατε και την τελευταία ιδέα που είπατε ότι θα πρέπει οι εταιρείε να δηλώνουν τα κέρδη τους σε κάθε χώρα. Τι ε, μπορείτε να το εξηγήσετε. Υποθέτω ότι είναι γιατί δεν μπορούμε να έχουμε μία εικόνα για τα παγκόσμια κέρδη. Οπότε τι προτείνετε να παίρνουμε ένα σταθερό ποσοστό σε κάθε χώρα για φόρο. Ποιος θέλει να μιλήσει πρώτος. Με την αντίστροφη σειρά προτείνω. Να ξεκινήσουμε από τον καθηγητή και ανάποδα από την πριν. Σας ευχαριστώ. Δημοσιεύσαμε μία έρευνα προσφάτως, ένα επιστημονικό μια επιστημονική εργασία. Θα προσπαθήσω να το συνοψίζω. Κοιτάξτε, το πρόβλημα με του υφιστάμενου κανόνες είναι ότι ε, δεν είναι σαφείς και επιτρέπουν στις αρχές ε, να φορολογήσουν τα κέρδη σε μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην ε, χώρα τους, αλλά πρέπει να την θεωρήσουν ανεξάρτητο τμήμα από τα άλλα κομμάτια της ίδιας πολυεθνικής, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Οπότε το BEPS ουσιαστικά απλά κρύβει τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Ειδικά όταν μιλάμε για το κόστος, μιλάμε για μια μεθοδολογία η οποία κατανέμει το κόστος π.χ. για τις κεντρικές υπηρεσίες. Αλλά για τα κέρδη δεν έχουν κάνει κάτι τέτοιο και έχουν κολλήσει στον κανόνα της απόστασης των λεγόμενων. Και βεβαίω τι γίνεται, υπάρχει ένας επαναχαρακτηρισμός των συναλλαγών. Π.χ. ξεκινάμε από την Google Ηνωμένου Βασιλείου και κοιτάμε αυτές τις συναλλαγές. Εγώ προτείνω ότι μπορούμε να έχουμε μια ενιαία προσέγγιση για να δούμε το παγκόσμιο κέρδος. Υπάρχουν δεδομένα, αρκεί να δούμε τους ισολογισμούς τους. Τους ενιαίους ισολογισμού που στέλνουν ε, στα χρηματιστήρια εντάξει, μπορεί να τα αλλάξουμε λίγο για φορολογικού σκοπού, αλλά γίνεται και το θέμα είναι μετά πώ κατανέμεται. Προφανώ για να πάμε σε μια κοινή φορολογική βάση ε, θα χρειαστεί μεγάλη προετοιμασία. Αλλά θα μπορούσαμε να κάνουμε μια κατανομή με βάση του ποια είναι τα παγκόσμια κέρδη και 25% θα πούμε ότι είναι λειτουργικό κόστος ή πωλήσει. Οπότε θα μπορούσαμε να έχουμε έναν ελάχιστο φόρο σε σχέση με τα συνολικά παγκόσμια κέρδη της εταιρεία ανάλογα με το κόστος και τις πωλήσει σε κάθε χώρα. Ναι, για το θέμα του πώς θα καταλήξουμε σε μια λύση για όλα αυτά. Κοιτάξτε, είχα εργαστεί για τον ΟΗΕ σε διάφορες εκστρατείες, σε διάφορες περιοχές. Δεν είμαστε βέβαια όλοι ήδη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλη φορολογική παράδειση, άλλη όχι. Όλοι μαζί πρέπει να τα βάλουμε με τους φορολογικούς παραδείσους και να δούμε τελικά ποιος είναι αυτός που μπλοκάρει τη διαδικασία με τον κώδικα δεοντολογίας και τις διαπραγματεύσεις ΩΣΑ, το πρόβλημά μου είναι ότι είναι απόρριτες. Δεν έχω δει κανένα κείμενο διαπραγματεύσεις πριν ληφθεί η απόφαση. Δεν ε, μπορούμε να επιβάλλουμε στις κυβερνήσεις να λογοδοτήσουν. Αυτό είναι το πρόβλημα και υπάρχει προηγούμενο και γι' αυτό εγώ ζητάω σε παγκόσμιο επίπεδο αποφάσεις και το ζητάω επειδή αυτό έγινε πριν από μερικά χρόνια κάποια στιγμή με πειρατεία όσον αφορά γενετικούς πόρους. Οι αναπτυσσόμενες χώρες κουράστηκαν τόσο πολύ να ακούνε ότι χάνουν δισεκατομμύρια δολάρια που άρχισαν να κλωτσάνε την ε, συνεργασία. Άμα δεν είσαστε διατεθειμένοι να μοιραστείτε τα κέρδη, δεν σας δίνω πρόσβαση στη χώρα μου. Έχει νόημα λοιπόν αυτό για χώρες που βλέπουν ότι δεν έχουν κέρδη. Μπορούν κάλλιστα να πούνε ότι δεν επιτρέπω την πρόσβαση της επιχείρησής σας στη χώρα μου. Εγώ θα στηρίξω τις δικές μου εγχώριες επιχειρήσεις. Φυσικά αυτή η κατάσταση πονάει όλους. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρξει σε παγκόσμιο επίπεδο συμφωνία. Και όταν λέμε ότι ο ΣΑ είναι πιο γρήγορος, δεν είμαι σίγουρη, γιατί τα τελευταία 50 χρόνια σπάνια κάποιος ε, βέβαια συντάσσει έγραφα τόσο γρήγορο όσο ο ΣΑ, αλλά δεν προχωράμε όσον αφορά τη λογοδοσία και την πολιτική βούληση. Οπότε, πού τη βλέπετε την ταχύτητα. Παγκόσμιες διαπραγματεύσεις πάντως δίνουν την ευκαιρία να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ναι, και εγώ θέλω να απαντήσω στην κυρία Γκόμες στην ερώτησή της για το απόρριτο. Είναι αλήθεια. Οι αναπτυγμένες χώρες δημιούργησαν τους φορολογικούς ε, παραδείσους που τους χρησιμοποίησαν βέβαια και Αφρικανοί ε, ηγέτες για τα δικά τους, τις δικές τους περιουσίες. Γκάνα, Κένια και άλλε αφρικανικές χώρες μπορεί κάλλιστα να είσαι φορολογικός παράδεισος, φορολογικό κέντρο. Είναι όμω ένα μοντέλο που εισάγαμε από τις ευρωπαϊκές χώρες. Οπότε την ευθύνη αναλογικά την έχουν περισσότερο οι ευρωπαϊκές χώρες. Εκείνες πρέπει να κάνουν περισσότερα θα έλεγα, αναλογικά. Οπότε το να λέμε ότι επειδή υπάρχουν κοινά συμφέροντα πρέπει και οι δύο πλευρές εξίσου, δεν στέκει. Μακάβαν, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, θα δώσω το λόγο στους εισηγητές. Από πλευρά της Αναπτυξιακής Επιτροπής, παρακαλώ, εσείς πρώτα πέντε λεφτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα αρχίσω λέγοντας ευχαριστώ για αυτήν την κοινή ακρόση. Είναι ζωτική σημασία να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα και από πλευράς ανάπτυξης. Μεγάλες ποσότητες χρημάτων με ένα κλικ μεταφέρονται από το ένα μέρος στο άλλο, οπότε σαφώς και πρέπει σε παγκόσμιο επίπεδο να έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία. Εγώ ήμουν υπεύθυνη λοιπόν για την έκθεση αυτή όσον αφορά τη φοροδιαφύγη και την φοροαποφυγή σε αναπτυσσόμενε χώρε και με αυτή την έκθεση ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει. Και θα αρχίσω με το εξή, για ο κύριο Μόμπα το είπε στην αρχή. Πόσο τεράστια είναι η κλίμακα του προβλήματος. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλάει για ε, ε δολάρια Στην έκθεση, λοιπόν, πιέζουμε, αλλά δυστυχώ όπως είπε και η Λίντα πριν, δεν εισακουστήκαμε στην Αδίσα Βέμπα για την, μετα... την αλλαγή της Επιτροπής ε, του ΟΗΕ σε κυβερνητική επιτροπή, ώστε οι χώρες να μπορούν εξίσου να συμμετέχουν στην δημιουργία των διεθνών κανόνων. Στον ΩΣΑ μόνο μια μικρή ομάδα πλούσιων χωρών κρυφά μέσα σε μια μικρή αίθουσα αποφασίζουν. Τα έγγραφα του Παναμά όμω δείχνουν για άλλη μια φορά ότι τα παγκόσμια προβλήματα πέτουν παγκόσμιε λύσεις. Και χρειαζόμαστε διαφάνεια. Οι αναπτυσσόμενε χώρες δεν συμμετείχαν στι διαπραγματεύσει BEPS εξίσου για να υπάρχουν διεθνείς κανόνες δεν μπορεί μόνο 34 πλούσιες χώρες να συμμετέχουν και να αποκλείονται 100 τόσες χώρες οι οποίες πλήττονται περισσότερο και να αποφασίζονται έτσι λύσεις για όλους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πρώτο βήμα που έχουμε κάνει. Ακολουθούμε λοιπόν το παράδειγμα κάποιων χωρών μελών για να υπάρξει αξιολόγηση και να αναλυθεί το θέμα των φορολογικών πολιτικών, πώς επηρεάζουν τα φορολογικά συστήματα των αναπτυσσόμενων χωρών και τα εισοδήματά τους. Και ήταν καλό που ακούσαμε νωρίτερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κ. Μεσεβίζη, ότι η Επιτροπή πιέζει τις χώρες μέλη για μια τέτοια αξιολόγηση. Επίσης, όταν διαπραγματευόμαστε συμφωνίες με τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες, λέμε ότι είναι καλύτερο να εφαρμόζουν το σύστημα του ΟΗΕ από εκείνο του ΟΣΑ. Κάποια από τα μέτρα που αποφασίζονται σε διεθνές επίπεδο είναι περιτά και συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, αλλά είναι άχρηστες για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Μπορεί να είναι καλά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν λέω, αλλά δεν φτάνουν κυρίως για να έχουμε ανάπτυξη. Αυτά τα μέτρα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαίτερες καταστάσεις και ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών. Η διαφάνεια ε, κοστίζει λίγο και αλλάζει την κατάσταση. Χρειαζόμαστε διαφάνεια λοιπόν να υπάρχει εμπιστοσύνη στα ΠΕΠΣ και σε αναπτυσσόμενες χώρες, την ανταλλαγή πληροφοριών με τις φορολογικές αρχές των χωρών αυτών, αλλά να λάβουμε υπόψη μας ότι χρειάζεται μια μεταβατική περίοδο για να αναπτύξουν τις ικανότητες που χρειάζονται για να συλλέξουν στοιχεία. Και δεν πρέπει κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο να αποκλείονται. Και έπειτα, μόνο ένα πλήρες CBCR μπορεί να βοηθήσει και να μην εκμεταλλεύονται οι πολυεθνικές το απόρριτο. Με την τωρινή πρόταση θα πρέπει να αποκαλύπτουν την κατάσταση και στην Αφρική και στην Αμερική. Μιλάμε για 750 εκατομμύρια. Αυτή είναι η απόφαση που σημαίνει 85 με 90% των πολυεθνικών να αποκλείονται με το όριο αυτό που βάλαμε για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Και η αναχώρα έκθεση τελικά δεν θα οδηγήσει σε τίποτα αν δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ δικαιοδοσιών. πολεμώνται βέβαια η ευρωπαϊκή φορολογική παράδειση, αλλά επιλεκτικά και καταλήγουμε σε έναν πολύ αδύναμο κατάλογο. Έχουμε πέντε λεφτά ακόμα, οπότε ολοκληρώστε παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος. Ναι, τα έγγραφα Παναμά κατέδειξαν ποια πρέπει να είναι η μερίσια διάταξη. Μην ξεχνάμε ότι δεν πρόκειται μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα χρήματα που χάνουν οι αναπτυσσόμενες χώρες κάθε χρόνο από τη χώρα αποφυγή έχουν σαν αποτέλεσμα να είναι αναποτελεσματικές οι δικές μας αναπτυξιακές πολιτικές. Γι' αυτό χρειάζονται γενικότερες λύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σάντζετ, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Αλλά θα σας τα πω στα ισπανικά, δεν έχετε αντίθεση. Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε που οργανώσατε αυτό το συμπόσιο, αυτή την κοινή συζήτηση. Ε, θεωρώ ότι από τα Panama Papers ανέκυψε το πόσα χρήματα κλέβουν κάποιοι άνθρωποι από τον κοινό κορβανά. Αλλά νομίζω ότι εμείς κάνουμε πολύ λίγα τον Ιούλιο. Όλες οι χώρες στην Ένωση, όπως πάντα, κάτι φτιάξαμε ένα κείμενο, το προσυπογράψαμε, αλλά δεν κάναμε τίποτα μετά. Και είχαμε το θεματολόγιο της Αντίσα τον Ιούλιο και είπαμε ότι όλοι θα πρέπει να ενδυναμώσουμε τη θωράκιση των εθνικών πόρων σε σχέση και με την ανάπτυξη, γιατί είπαμε ότι είναι κάτι το πάρα πολύ βασικό, ούτω ώστε να υπάρχουν περισσότεροι πόροι για την ανάπτυξη. Εγώ προσωπικά ε, θεωρώ ότι ε, έχουμε τα εξή δήματα που αναδύονται. Υπάρχουν κάποιε κοινέ αξίε, όπω η κοινωνική δικαιοσύνη, γιατί ακριβώ μέσω τη δίκαιες φορολόγησης, έχουμε αναδιανεμητικά συστήματα και έτσι μπορούμε να, αυξάσουμε, να αυξήσουμε τους ε, πόρους ε, και έτσι μπορούμε να έχουμε περισσότερη κοινωνική συνοχή, να καποτεμήσουμε τις ανισότητες, τις κοινωνικές των ε, δύο φύλων και έχουμε και τους ε, στόχους του ΟΗΕ που για το 2030. Αν καταπολεμήσουμε την ανισότητα θα έχουμε περισσότερη συνοχή. Έτσι ενισχύουμε τον εκδημοκρατισμό και την ιδιότητα του πολίτη. Επίσης θα πρέπει στους εσωτερικούς πόρους να δούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει δημοκρατία αλλά και διαφάνεια. Θα πρέπει να εκδημοκραστεί η οικονομία και να εξυπηρετεί τον κόσμο και όχι το αντίθετο. Όταν δεν υπάρχει διαφάνεια για τις ροές κεφαλαίων, ε, τότε οδηγούμε σε σημαίνει κατάσταση όπου αυτό είναι σε τραγική κατάσταση και άρα χρειάζονται έλεγχοι πολλές φορές ε, κατά της φοροαποφυγής ε, γιατί πολλές φορές το ξέρουν πόρων σημαίνει ότι ενισχύονται εγκληματικές οργανώσεις και αυτό στέφεται κατά του κόσμου η λίστα Φαλσιανή τα Panama Papers λοιπόν έκαναν θόρυβο, αλλά δεν έγιναν πολλά πράγματα. Ε, πατρίδα των εγκληματιών είναι μόνο το χρήμα. Αλλά πρέπει να υπάρχουν κάποιε πολιτικέ, επίγοντα μέτρα που να θέσουν τέρμα σε τέτοιε πρακτικέ. Ε, Επομένω να υπάρχουν περισσότερε εκθέσει, περισσότερο αυτό το reporting αναχώρα, ε, αναθεώρηση του φορολογικού δικαίου και εκμετάλλευση των επενδυτικών και εμπορικών συμφωνιών που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Θα πρέπει όμως να υπάρχει και ποινικό δίκαιο που να προβλέπει αυτά τα εγκλήματα που καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν θα πρέπει ούτε μία μέρα παραπάνω να μείνουμε αδρανείς. Καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα πρέπει με αυτού του είδους την φορολογική πειρατεία να δούμε πόσο ε, στρέφονται αυτά τα εγκλήματα κατά των εμπισόμενων χωρών γιατί χρειάζεται δικαιοσύνη για να πρετανεύσει η κοινή λογική. Να κάνουμε ό,τι πρέπει από το χέρι μας, ούτως ώστε να σταματήσει να υπάρχει ατιμορρησία σε σχέση με αυτά τα φαινόμενα. Η κυρία Μακάβαν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τις δύο. Συνοψίσατε πάρα πολύ εύστοχα όλα τα θέματα. κ. Λαμασούρ λέει να τον ε, συμπαθείτε γιατί λόγω της απεργίας στη Γαλλία έπρεπε να φύγει επιγόντως για να προλάβει. Οπότε αναδείχθηκαν δηλαδή, πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα και μας είπατε επίσης τι γίνεται με το σύστημα του ΟΗΕ. Και ελπίζω η Επιτροπή μας να προλάβει υπόψη. και είπαμε ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε και με την ε, Αφρικανική Ένωση. Και αυτό αφορά και την Επιτροπή που αντιπροσωπεύεται, προσωπείται τέλο στην αίθουσα. Κάτι πρέπει να γίνει για αυτέ τι πρακτικέ, αλλά συγκεκριμένα ζητήματα ήταν αυτό το οποίο είπατε για το ότι τα έξοδα, τα φορολογικά έσοδα μάλλον τα οποία δεν μπορεί να εισπραχθούν από μία πολυεθνική είναι σαν όλο τον προπολισμό παιδεία τη Ζάμπη. Θυμάμαι για τον έμπολα, για τη Λιβερία. Λέγαμε ότι όλο το μπάτζετ είναι λιγότερο από το όσα χρήματα δαπανώνται στην πόλη μου και μιλάμε για μία χώρα και για ένα χρόνο εξόδων για το έμπολα. Δεν είναι να παραμελούμε αυτά τα φορολογικά προβλήματα. Δεν θέλω να γίνεται αιμοδοσία προς χώρες της Αφρικής. Θέλω οι χώρες οι ίδιες να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους με τα δικά τους έξοδα. Όλοι λένε για την μετανάστευση, με τις αιτίε της μετανάστευσης, να κάνουμε το α, το β. Αλλά να, ποια είναι η αιτία. Φτώχεια, δεν υπάρχουν κρατικές υπηρεσίες, η κοινωνία είναι διαλυμένη, γι' αυτό και είμαι ευγνώμων προς την ε, Επιτροπή των Φορολογικών Ρυθμίσεων. Έτσι θα πετύχουμε τους στόχους τους αναπτυξιακούς και πάλι ευχαριστούμε όλους. Βιώσαμε πάρα πολύ από το χρόνο και είχαμε πάρα πολλά να πούμε. Αλλά μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας να οργανώσετε και ό,τι θέλετε. Ευχαριστούμε και του διερμήνες για τον έξτρα χρόνο που μας αφιέρωσαν.